Um, Καλό απόγευμα σε όλους και όλες. Αν μπορείτε να καθίσετε λοιπόν μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Το πρώτο θέμα στην ημερησία διάταξη είναι η έγκριση αυτής της ιδίας ημερησίας διάταξης. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μπορώ να θεωρήσω ότι έχει εγκριθεί. Δεύτερο θέμα στην ημερησία διάταξη είναι οι ανακοινώσεις της Προέδρου οι οποίες είναι αχρίαστες, δεν έχω καθόλου. Και μπορούμε να περάσουμε τώρα στο τρίτο θέμα. Κεφαλαιακές απαιτήσει το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και τις πράξεις επαρτιτλοποίησης καθώς και τον υποπτικό έλεγχο των μισθολογικών πολιτικών. Εδώ εξετάζουμε τις τροπολογίες και δίνω αμέσω το λόγο στην εισηγήτριά μας την Αρλέν Μακ Ευχαριστώ, <clears throat> Σάρων. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους οι οποίοι χρησιμοποίησαν το χρόνο να καταθέσουν τροπολογίες, πολλές από τις οποίες νομίζω ότι βελτιώνουν το κείμενο και θα συναντηθώ προσωπικά όλους αυτούς που κατέθεσαν τροπολογίες και φυσικά και τους σκιώδεις εισηγητές έχουμε διερμηνία εδώ. Έχουμε πρόβλημα με την μετάφραση προς τα γερμανικά. Ακούτε τα γερμανικά. Εντάξει, ακούγονται καλά τα γερμανικά. Αυτό το οποίο θα ήθελα να κάνω σήμερα είναι το εξής. <clears throat> Υπήρξε η πρόταση να αναβάλουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να την κάνουμε σήμερα την ανταλλαγή απόψεων για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε λιγάκι στο να εξετάσουμε τις τροπολογίες και να καταλήξουμε σε κάποιες συμβαστικές λύσεις. Σίγουρα θα μπορέσουμε να βρούμε κάποιες συμβαστικές λύσεις γιατί οι τροπολογίες είναι πολύ χρήσιμες οι περισσότερες από αυτές και συμπληρώνω αυτές που κατέθεσα εγώ η ίδια, αλλά θέλω να ενημερώσω τους συναδέρφους σε σχέση με τις συζητήσεις που έχουν γίνει στην Επιτροπή Βασιλείας στην Ιαπωνία, που μας δίνουν και μια νέα προοπτική στο έργο μας. Να σας πω λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι ότι οι τροπολογίες όπως τις έχω δει μπορώ να τις κατατάξω σε τέσσερις κατηγορίες. Πρώτον, <clears throat> αυτές οι οποίες αντικατοπτρίζουν την άσκηση πίεσης από τον τραπεζικό τομέα για να καθυστερήσουν την εφαρμογή των κανόνων για κεφαλαιακή επάρκεια και να εξαιρέσουν ορισμένε κατηγορίε κεφαλαίων. Η δεύτερη κατηγορία έχει να κάνει με τι αμοιβέ των στελεχών. Και αυτό το οποίο βρίσκω πολύ θετικό σε αυτέ τι τροπολογίε είναι ότι αναγνωρίζουν την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε του κινδύνου οι οποίοι ελοχεύουν στι πρακτικέ αμοιβή των στελεχών που έχουμε στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο ουσιαστικά και χαιρετίζω το γεγονό ότι όλοι αυτοί που κατέθεσαν τροπολογίε συμμερίζονται και τι δικέ μου τι ίδιε ανησυχίε που παρουσιάζονται στις δικές μου τροπολογίες. Λοιπόν, είναι συμπληρωματικές αυτές οι τροπολογίες με τη δική μου, τις δικές μου που εγώ προσπαθώ να εδραιώσω τις αρχές που εγκρίνανε οι G20. Τονίζουν ορισμένοι ότι πρέπει να σπάσουμε την σύνδεση μεταξύ της κουλτούρας των πόνους και των υπερβολικών ρηψοκίνδυνων ενεργειών για αυτό το στόχο. Εγώ κατέθεσα ως τροπολογίε που έχουν να κάνουν με την εμπλοκή των επενδυτών και των ε, μετόχων, ώστε να υπάρξει μια επιτροπή για τις αποδοχές που να ελέγχει τα μπόνους και να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και επίσης μια ψηφοφορία των μετόχων ώστε να υπάρξει ένας διαχωρισμός των κερδών μεταξύ των διακρατούμενων κερδών και των κερδών που διανέμονται σε μερίσματα και μπόνους. Όλα αυτά για να μπορέσουμε να έχουμε μια σωστή ισορροπία μεταξύ των διακρατούμενων κεφαλαίων και των μπόνους και των μερισμάτων και φυσικά να εξετάσουμε όλη την πολιτική αποδοχών. <clears throat> Αλλά θα ήθελα να δω πώς μπορούμε να έχουμε κάποιες συμβαστικές τροπολογίες για τα θέματα αποδοχών. Πολλές από τις τροπολογίες που έχουν κατευθεί από τους συναδέλφους μου νομίζω ότι βελτιώνουν το κείμενο. Τρίτος χώρος τροπολογιών αφορά τα ειδικά εποπτικά μέτρα για πολύπλοκες επανατιτλοποιήσεις και νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε μια συμβαστική θέση επί τη βάση αυτών των τροπολογιών, ιδίω για κάποιες από τροπολογίες που ζητούν να υπάρξει και περισσότερη δουλειά από την Κομισιόν για την ανάλυση της αγοράς επανατιτλοποίησης Και εδώ το ερώτημα είναι αν θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την δέουσα επιμέλεια στον τομέα αυτό πολλοί από του ε, ρυθμιστέ είπαν ότι δεν έχουν την ικανότητα να εξασφαλίσουν πλήρω την εποπτεία του τομέα αυτού. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι απαιτείται από την πλευρά μια πλήρου ρυθμιστική εποπτείας. Τέταρτο στοιχείο είναι ο δημοκρατικό έλεγχο. Και πάλι βρίσκω πάρα πολύ θετικέ τροπολογίε, μερικέ είναι πάρα πολύ τεχνικέ. Θα μπορώ να συζητήσω με τα, ε, με τα μέλη τη Επιτροπή μα. Νομίζω ότι μπορούμε να τι ενσωματώσουμε αλλά θέλω να σταθώ στο κύριο θέμα, που είναι το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Θα ξέρετε ότι υπήρξε μια συνάντηση στην Ιαπωνία στις 9 Απριλίου της Επιτροπής Βασιλείας και στη συνάντηση αυτή τόνισαν ορισμένα κράτη ότι είχαν προβλήματα με την ε, ε, ημερομηνία εφαρμογής και θέλουν μόνο σταδιακά να εφαρμοστούν οι απαιτήσει της οδηγίας για την κεφαλαιοϊκή επάρκεια 3. Νομίζω λοιπόν ότι είναι χρήσιμο να δούμε ποιο είναι ο αντίκτυπο αυτών των μέτρων. Δεν μπορούν οι τράπεζε να έρχονται και να λένε να καθυστερήσουμε επειδή έτσι θέλουμε και θέλουμε καθυστέρηση. Αλλά αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να λάβουμε υπόψη μα το γεγονό ότι η ίδια η Επίτροπη τη Βασιλεία αλλάζει την άποψή τη σε ορισμένα μέτρα. Λέει ότι θέλει να αναθεωρήσει ορισμένα μέτρα. Επομένως αυτό μπορεί να είναι ένα επιχείρημα όχι για καθυστέρηση αλλά για μια σταδιακή εφαρμογή ορισμένων απαιτήσεων και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι λογικό να το ενσωματώσουμε και στο δικό μας χρονοδιάγραμμα. Και θα έχουμε στα μέσα Μαΐου μια έκθεση αντικτύπου, νέες προτάσεις τον Ιούνιο. Όλα αυτά δεν πρέπει να καθυστερήσουν φυσικά το έργο το οποίο κάνουμε εμείς για την έκθεση αυτή, αλλά πρέπει να τα λάβουμε αυτά υπόψη καθώς συντάσσουμε τις τροπολογίες ε, συμβιβασμού και φυσικά θα ακούσουμε και τις απόψεις των σκιωδών εισηγητών και του, της Προέδρου για το ποια είναι η πιο πρόσφορη χρονική στιγμή για την ε, τελική ψηφοφορία. Αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε, να συνεχίσουμε την πρόοδο, αγαπητοί συνάδελφοι. Η οδηγία αυτή <clears throat> θα πρέπει να εγκριθεί πριν από το τέλος του χρόνου. Χρειαζόμαστε νέες ρυθμίσεις πριν από το 2011. Ελπίζω ότι θα υπάρξει αυτή η υποστήριξη από όλους για να μπορέσουμε να έχουμε το ταχύτερο δυνατόν αυτές τις νέες προτάσεις. Και απλώς για το θέμα της λεγόμενης πατρογονικής ρήτρα, ιδίως για την επανατητοποίηση του grandfathering. Νομίζω ότι εμείς ως ε, νομοθέτες δεν πρέπει να υποστηρίξουμε μια υπερβολικά ευρεία πρόταση πατρογονικής ρήτρας, grandfathering, γιατί αυτό μπορεί να αφήσει κάποια τοξικά στοιχεία ενεργητικού στον ισολογισμό τραπεζών που δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τις απώλειες, επομένως ο ρόλος της Επιτροπής μας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι σε αυτή την περίπτωση να μην αφήσουμε τον φορολογούμενο έκθετο σε μια περαιτέρω ενέργεια διάσωσης. Δεν πρέπει λοιπόν να θεωρήσουμε ότι είμαστε σε μια κατάσταση όπου δεν κινδυνεύουμε πια να επαναληφθεί η χρηματοοικονομική κρίση και γι' αυτό είναι απαραίτητο να εργαστούμε με τις τράπεζες και να τις πείσουμε να έχουν ε, αποθέματα κεφαλαίου για να καλύψουν όλους τους κινδύνους ξέρω ότι θα πιεστούν για να μπορέσουν να επιτύχουν την κεφαλαιακή επάρκεια η οποία χρειάζεται. Χρειάζεται όμως να τους πείσουμε τις τράπεζες και να τους δώσουμε τα κίνητρα για να τα πετύχουν αυτά. Και θέλω να υπενθυμίσω ότι οι ορισμένε τράπεζε ζήτησαν ενεργά να υπάρχει καθυστέρηση, αλλά είναι οι ίδιε τράπεζε οι οποίε δίνουν υπερβολικά μπόνου στα στελέχη του. Επομένω, μήπω θα πρέπει κάποια από αυτά τα χρήματα να τα χρησιμοποιήσουν για να έχουν κεφάλαιο αποθεματικό και όχι να πληρώνουν τεράστια μπόνους όπως έγινε στο τέλος του 2009, αρχές 2010. Προτείνω λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι να δούμε το πώς τροποποιούνται οι διατάξεις της ε, Βασιλείας. Θα πρέπει να βρούμε ένα επικοδομητικό τρόπο για να μπορέσουμε να πείσουμε τις τράπεζες να καλύψουν τις απαιτήσει του CRD3, της οδηγίας δηλαδή για την κεφαλαιακή επάρκεια 3, αλλά δεν θέλουμε η Επιτροπή μας να οδηγήσει σε κινδύνους για το φορολογούμενο, και συγχρόνως θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει και κάποια δυνατότητα να συναντηθούμε όλοι και εγώ και οι σκιώδεις πολλοί από τους οποίους δεν μπόρεσαν να έρθουν στο Στρασβούργο, αλλά επειδή η Επιτροπή της Βασιλείας θα πάρει και νέες αποφάσεις στην Ιαπωνία, θα είναι χρήσιμο να συνεκτιμήσουμε όλα αυτά τα στοιχεία, χωρίς όμως να καθυστερήσουμε αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε αυτά τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή και να διτηρήσουμε ακόμα την πορεία μας για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι πλήρω την 1η Ιανουαρίου του 2011, εφόσον το θέλει και ο Θεό. Και θα ήθελα να έχω και τι απόψει όλων των συναδέλφων για το θέμα αυτό. Μέχρι στιγμή έχουν κατατεθεί 227 τροπολογίε, είναι πολυθετικέ πιστεύω και ελπίζω θα μπορέσουμε να βρούμε επωφελεί συμβιβαστικέ λύσει για να βελτιώσουμε το κείμενο. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριο Καρά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να πω καταρχήν ότι είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση μεταξύ των σκιωδών εισηγητών και της εισηγήτριας για το θέμα αυτό. Σε σχέση με τις τροπολογίες, δεν έχουμε ακόμα διατυπώσει πλήρως τις ε, ενδεχόμενες συμβιβαστικές τροπολογίες, αλλά έχουμε προχωρήσει στο θέμα αυτό. Το δεύτερο που θέλω να τονίσω είναι ότι συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι από τη μία πλευρά δεν πρέπει να καθυστερήσουμε ιδιαίτερα, αλλά Συγχρόνως, δεν πρέπει να προχωρήσουμε μόνοι μας ως Ευρώπη τη στιγμή που αυτό θα οδηγήσει σε δυσκολίες μέσα στην Επιτροπή της Βασιλείας. Θα πρέπει να παραμείνουμε μέσα στο σωστό χρονοδιάγραμμα, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσαμε να αναβάλουμε την ε, ψηφοφορία για την επόμενη εβδομάδα και αυτό δεν θα καθυστερήσει το χρονοδιάγραμμα μέχρι το καλοκαίρι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά προβλήματα ακόμα στο, πλαίσιο της Επιτροπής ε, της Βασιλείας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπουμε ότι δεν είναι έτοιμες οι Ηνωμένες Πολιτείες να εφαρμόσουν μια σειρά από ρυθμίσεις της Επιτροπής της Βασιλείας μέχρι τα μέσα, πριν από τα μέσα του 2011 και θα ήταν απαραίτητο να καταλήξουμε και σε μια κοινή στάση σε διαβουλεύσει με τους εταίρους μας από τις άλλες χώρες του κόσμου σε σχέση με την εφαρμογή των αποφάσεων της Βασιλείας. Είναι επίσης απαραίτητο να δώσουμε ένα πολιτικό μήνυμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να τονίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να εφαρμόσει τις αποφάσεις των G20 και γι' αυτό το λόγο δεν θα πρέπει να αφήσουμε να υπάρχει να πλάνεται καμία αμφιβολία ότι εμεί είμαστε έτοιμοι για την ταχύτερη δυνατή εφαρμογή των αποφάσεων σε σχέση με τις αμοιβέ των στελεχών των τραπεζών. Ίσως αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί χωριστά, όπως είπε η η Για μένα πάντως είναι λογικό να ψηφίσουμε τον Ιούνιο στην Επιτροπή μας και για μας είναι σε επίπεδο περιεχόμενο τα εξής. Ότι πρώτα η Κομισιόν θα πρέπει να <clears throat> αντιμετωπίσει το ταχύτερο δυνατό τα εκκρεμή θέματα τα οποία υπάρχουν και εδώ υπάρχουν σε σχέση με το, με το CRD2, δηλαδή την κεφαλουχική, οδηγία κεφαλουχικής επάρκειας υπαριθμών 2, είναι επαρκειας παριθμων 2 ειναι απαραιτητο να εξασφαλιστεί κάποιο συντονισμός και σε παγκόσμιο επίπεδο και προς το παρόν δεν έχουμε την αντίδραση της Κομισιόν σε σχέση με τα θέματα αυτά ε, και αυτό αφορά ιδίω τα θέματα τίτλοποίησης. Είχαμε τονίσει εμείς ότι η Κομισιόν θα πρέπει να ελέγξει στα πλαίσια της δεύτερης οδηγίας για την κεφαλουργική επάρκεια να εξετάσει μία αύξηση του ποσοστού ασφαλείας ώστε να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις στην αγορά τιτλοποίησης δεν πρέπει να καθυστερήσουμε ιδιαίτερα τη μετάβαση από τη Βασιλεία 1 στη Βασιλεία 2. Μια γενική ρήτρα αναθεώρησης για την πολιτική αποδοχών θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι η Ευρώπη θα μπορέσει να παραμείνει ανταγωνιστική και η συμμετοχή των ευρωπαϊκών ε, αρχών εποπτείας τράπεζας και εποπτείας αγοράς <clears throat> νομίζω ότι είναι απαραίτητη και το θέμα των πολυπλόκων πράξεων επατοτοποίησης είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και θα πρέπει σε αυτά ενδεχομένως να καθυστερήσει η ψηφοφορία, αλλά είναι απαραίτητο να μπορούμε να έχουμε μια σαφή πολιτική σε ό,τι αφορά τις αποδοχές. Νομίζω ότι η Κομισιόν θα πρέπει να δώσει στην Επιτροπή μας το ταχύτερο δυνατό απαντήσει σε όλα τα εκκρεμή θέματα που αφορούν την οδηγία κεφαλουχική επάρκεια υπαριθμών 2, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατό. Ευχαριστώ. Οι σκιώδει θέλουν να μιλήσουν, Βίκη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Αρλίν, για τη δουλειά που κάνεις και ήταν πολύ χρήσιμε οι συνεδριάσει των σκιωδών εισηγητών και περιμένουμε και την επόμενη συνάντησή μα αυτήν την εβδομάδα, όπω είπα και στην προηγούμενη ανταλλαγή απόψεων. Είναι απίστευτα σημαντικό νομοθέτημα αυτό, διότι είναι συγκεκριμένη δράση που περιμένουμε να αναλάβουν οι τράπεζε τώρα και να ξεκαθαρίσουν ε, το όλο μπέρδεμα που υπάρχει στον αφορά τις ενέργειέ του, τι οικονομικέ και ε, κυρίως την πολιτική αμοιβών που ακολουθούσαν, τη φοβερή διάφορες τράπεζες. Σε προηγούμενες ακράσεις, είπα ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνουν πράγματα και θα πρέπει η σορευτική συνέπεια του αυξανόμενου κεφαλαίου που ζητάμε όχι μόνο στο CRD3 αλλά και στο CRD4 να μην θέσει τροχοπέδι στο κεφάλαιο το διαθέσιμο για δανειοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Πότε ξεκινάμε είναι το θέμα την εφαρμογή των μέτρων και ποιος θα είναι ο αντίκτυπος. Και πώς θα εφαρμοστεί σε παγκόσμιο επίπεδο και θα συμφωνηθεί όχι μόνο σε ευρωπαϊκό. Απ' τη μία είμαι ευχαριστημένη που άκουσα ότι η συγγήτρια προτείνει να εξετάσουμε τι έγινε στην προηγούμενη συνεδρίαση της Βασιλείας, της ομάδας Βασιλείας. Ήταν θετικό θεώρησα ότι είπα, είπαν ότι θα μπορούσαν να ξεκινήσουν να εφαρμόσουν τα μέτρα από τα μέσα του επομένου έτου. Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι φορείς εποπτείας του Ηνωμένου Βασιλείου εξακολουθούν να θέλουν εφαρμοστεί από 1η Πρώτου του 2011. Στην πρώτη μας προθεσμία δηλαδή. Άλλες τράπεζες όμως πίεζαν για παρατάσεις πολύ μεγαλύτερες μέχρι το 2014. Κάποια μέλη τη επιτροπή πρότειναν τέτοια παράταση. Εγώ πιστεύω ότι είναι κάτι απαράδεκτο αυτό. Πέντε χρόνια μετά από αυτή τη χρηματοστική κρίση να μην έχουμε ξεκαθαρίσει ακόμα ε, τι γίνει και όσον αφορά το κεφάλαιο που αντιστοιχούσε στην ιστορική επανατιτλοποίηση. Υπάρχουν στοιχεία από την ομάδα Βασιλείας, συνεδρίασαν, συζήτησαν το θέμα την περασμένη εβδομάδα πρέπει να περιμένουμε μέχρι μέσα Μαΐου να εξετάσουμε αυτά τα αποτελέσματα και θέλω να δω πώς θα έχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες. Χρειάζεται κάποια δημοσιότηση όσον αφορά τα στοιχεία, τους αριθμούς. Χρειάζεται διαφάνεια όσον αφορά τα στοιχεία που εξετάζονται. Δεν αρκεί οι τράπεζες να λένε δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό γιατί θα έχει μεγάλο αντίκτυπο χωρίς να μπορούμε να το επαληθεύσουμε αυτό. Τώρα, Βάσει ποιων στοιχείων ενεργητικού. Θα ήθελα να ξέρω ακριβώς που έγκυται το πρόβλημα στον αφορά τη διατύπωση. Γι' αυτό υπέβαλα σχετικά δύο τροπολογίες. Η μία είναι τεχνικής φύσης. για συνθετικά δομημένες τιτλοποιήσεις που είναι στοιχεία ενεργητικού που προχρονολογούνται της κρίσεως. Και μέγιστα όρια απώλειας όσον αφορά τα παράγωγα στοιχείων ενεργητικού. Ακολούθησα τη διατύπωση όσον αφορά το σχετισμό που θα μπορούσε ε, να συμπεριληφθεί όσον αφορά το ανώτατο όριο απολειών. Εγώ δεν θέλω να καθυστερήσει η εφαρμογή για όλα τα ιστορικά στοιχεία ενεργητικού. δίνουμε πολύ χρόνο έτσι στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κυρίως αν η προθεσμία είναι μετά το 2014. Η διατύπωση για τις αμοιβέ, για τις αποδοχές, ίσως εκεί μπορούμε να πετύχουμε κάποιο συμβιβασμό. Ίσως το κείμενο που συμφώνησαν οι G20. Αν καταφέρουμε συμβιβασμό μέχρι το τέλος του έτους θα είναι πολύ επικοδομητικό. Εγώ ανησυχώ λίγο. Οι τράπεζε των ΗΠΑ πληρώνουν τι αμοιβέ πριν τα Χριστούγεννα και οι ευρωπαϊκέ τράπεζε μετά τα Χριστούγεννα. Καταβάλουν τα μπόνους. αν θεσπίσουμε νομοθεσία στο ενδιάμεσο, κάποιοι θα προσπαθήσουν να πληρώσουν πιο γρήγορα για να αποφύγουν την εφαρμογή της νομοθεσίας. Μπορούμε να το συζητήσουμε για να δούμε πώς μπορούμε να το ελέγξουμε. Πρέπει οι τράπεζες να ξεκινήσουν να δρουν τώρα. Χρειάζεται διαφάνεια όσον αφορά τα στοιχεία. Και είναι απαράδεκτο ότι κάποιε κυβερνήσει και κάποιε τράπεζε λένε αναβάλλετε, αναβάλλετε, αναβάλλετε, διότι δεν θέλουμε να αποκολύψουμε τα επίπεδα στοιχείων ενεργητικού που έχουμε όσον αφορά την έξοδό μα από αυτή την περίοδο ε, των τοξικών παραγόγων. Κυρία Κάμπερ, όχι κύριος, ο κύριος Κανφίνα. Δεν θα παρουσιάσω τις τροπολογίες μία-μία γιατί θα τις ξανασυζητήσουμε, αλλά για τις προθεσμίες. Υπάρχει το θέμα της διεθνούς συνεργασίας και της ανάγκης για συνέπεια των διεθνών κανόνων, αλλά επίσης και το μήνυμα που θα στείλουμε στους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο γιατί και ο τύπος αναμένει κάτι που να δείχνει ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές ξανάρχισαν να λειτουργούν. Συγγνώμη, there is no translation. Ακούγονται τα γερμανικά στο αγγλικό κανάλι. Ναι, πολύ δύσκολα. Πέστε κάτι να δούμε αν μεταφράζουν. Α, να ξαναρχίσετε, να ξαναρχίσετε. Έλεγα λοιπόν ότι για το χρονοδιάγραμμα τρία θέματα τίθενται. Πρώτον, θέλουμε διεθνή συνεργασία και συνεργασία με τη ΣΥΠΑ, αλλά επίσης δεν θέλουμε να νομίσουν οι πολίτες ότι υπάρχει υπαναχώρηση και καθυστέρηση της εφαρμογής των νέων κανόνων, ιδιαίτερα για τις απολαβές ή για την απόδοση των κεφαλαίων, εφόσον μάλιστα ο τύπος δείχνει ότι ξανάρχισαν τα ίδια τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Έχει μια ευθύνη εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποδείξει, να δείξει ότι ο Ευρωπαίος νομοθέτης και η νομοθέτρια είναι ενεργοί γιατί θέλουμε να φανεί ότι οι κανόνες αυτοί θεσπίζονται όχι μόνο για λόγους πολιτικούς και ηθικούς αλλά και για να μην ξαναυπάρξει η ίδια διατάραξη του συστήματος. Τεχνικά λοιπόν καταλαβαίνω ότι χρειάζεται κάποιος χρόνος για να προσαρμοστούμε στους νέους κανόνες αλλά όσο περισσότερο περιμένουμε και καθυστερούμε τόσο περισσότερο θα φαίνεται ότι πολιτικά, αν φτάσουμε στο 14 και 15, οι πολίτες θα αρχίσουν να διαμαρτύρονται. Έξι χρόνια μετά την κρίση εφαρμόζονται οι κανόνες. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αν περιμένουμε πέντε χρόνια μέχρι να εφαρμοστούν οι κανόνες θα προλάβει να ξεσπάσει καινούργια κρίση. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρουμε επίσης ότι η πίεση των τραπεζών και το lobbying έχουν πάντοτε αντιρρήσεις. Πότε οι κεφαλαιακές απαιτήσει αγνοούν το ένα, πότε το αένα αγνοεί τις κεφαλαιακές απαιτήσει. Και κάθε φορά ζητούν αναβολή. Ε, πρέπει να σφυρίξουμε το πέρας του αγώνα. Το πέρας του διαλύματος μάλλον. για να μην φανεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι σε θέση να νομοθετήσει, ιδιαίτερα για τις αποδόσεις. Για να δούμε τώρα. Όλοι σημαίνει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Σμίτ δηλαδή. Θα πω κάτι που ίσως να μην το εκτιμήσουν όλοι. Οι τράπεζες είναι πολύ σημαντικές για την ε, οικονομία της αγοράς, ακόμη και για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς. Είναι περίεργο που χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους ορολογία εδώ και ρητορία. Στις δικές μου τουλάχιστον τροπολογίε και σε άλλες θέλουμε την ε, αναδόμηση της οικονομίας στην Ευρώπη που έχει ζημιωθεί πολύ από την κρίση. Και αν θέλουμε να επιδείξουμε φρόνηση, δεν πρέπει να τα κάνουμε τα πράγματα πρόχειρα και βιαστικά. Για να μην αυξηθούν ακόμη οι ζημίες που υπέστησαν ορισμένοι. Να έχουμε λοιπόν εξισορροπημένη στάση. Ε, και μένα με έχουν πιέσει τράπεζες. Γιατί αν πούμε ότι καμία τράπεζα δεν έχει επαρκή κεφάλαια, αυτό είναι λάθος. Μερικές τράπεζες που θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα με τη νέα οδηγία δεν έχουν πρόβλημα έλλειψης κεφαλαίων, έχουν προβλήματα όμως άλλα από το νέο σύστημα θα έχουν. Και γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα που Μπορείτε να δεχτείτε κυρία Μακάρθη το facing in, την προοδευτική εφαρμογή δηλαδή. Δεν πρέπει να ντρεπόμαστε γι' αυτό ή να λέμε ότι δεν ε, δίνουμε σωστό μήνυμα στους πολίτες και το κοινό ή οποιουσδήποτε είπατε προηγουμένως ορισμένοι. Γιατί ένας από τους στόχους μας εδώ στην Επιτροπή είναι να ακούσουμε ή τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να ακούσουμε διαφορετικές απόψεις με τρόπο ρεαλιστικό όμως. Έτσι γίνεται και στα παραμύθια που διάβαζα και εγώ στα παιδιά μου. Όταν φοβόνταν, μου τους έλεγα «Μα μη στεναχωριέστε, στο τέλος θα πάνε όλα καλά». Και μια από τις σημαντικότερες οδηγίες που έχουμε να εξετάσουμε είναι αυτή που έχουμε σήμερα. Δηλαδή, για μένα, για μένα, οι τελικές σφαιρικές επιπτώσεις είναι το σημαντικότερο. Και πρέπει να δούμε τι γίνεται και σε άλλες υπήρους. The North Atlantic. Ιδιαίτερα εννοώ τις σχέσεις μας με τις χώρες του Βορείου Ατλαντικού από την άλλη μεριά όμως του ωκεανού. Την άλλη από πίσω. Και Φαντάζομαι ότι δεν θα δεχτεί η συγγήτρια όλες μου τις τροπολογίες, αλλά τουλάχιστον μερικές να δεχτεί, μερικές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την συγγήτρια. Κάποιες παρατηρήσεις μόναχα θέλω να κάνω. Υπάρχουν πολλά πράγματα πρέπει να κάνουμε σε σχέση με τις κεφαλαιοχικές, τα θέματα κεφαλαιοχικής επάρκειας. Αλλά αυτά πρέπει να τα δούμε σε διάφορα επίπεδα. Στο επίπεδο της ε, Βασιλείας, στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά επίσης αυτά πρέπει να τύχουν συζήτηση και σε εθνικό επίπεδο. Άμα δω μοναχά την πρόταση της εισηγητρίας, την ποιότητα της ε, πρότασης, Τη Κομισιόν μάλλον, όχι της νομίζω ότι υπάρχει μια σώρευση μέτρων που θα μπορούσε να υπερβαρύνει, να δημιουργήσει υπερβολικό άχθος για τις τράπεζες και τα πιστοτικά ιδρύματα. Η πρόταση για το CRD3, εδώ είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε καταρχήν ε, να μια ισότητα ανταγωνισμού. Επομένως, θα πρέπει να αντιστοιχεί η πρόταση για το CRD3 με τις ε, ρυθμίσεις της ε, Βασιλείας. Η μεγαλύτερη μου ανησυχία και το σημείο που είμαι πιο επικριτικός είναι ότι η ημερομηνία εφαρμογής αναφέρεται ως Δεκέμβριο του 2010. Εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς και είναι πραγματικά μη ρεαλιστική μια τέτοια εφαρμογή. Όλοι ξέρουμε ότι είναι απαραίτητα αυτά τα μέτρα, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία μεταξύ μας, αλλά δεν θα βοηθήσει να λειτουργήσουμε σε βεβαιασμένο, τρόπο για την εφαρμογή αυτό το μέτρο, γιατί αυτό μπορεί να αποδειχθεί και αντιπαραγωγικό. Λοιπόν, πιστεύουν πολλοί ότι, ότι από τη στιγμή που έχουμε μια κρίση πολλαπλασιάζονται οι απαιτήσει για τις τράπεζες και πολλές φορές δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν σε αυτές τις ανάγκες. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια νέα χρηματοοικονομική κρίση που φοβόμαστε όλοι αν προκύψει. Και επίσης υπάρχουν άλλα στοιχεία στην έκθεση της κυρίας Μακάρτη τα οποία εγώ τα υπογραμμίζω. Και εξάλλου υπογραμμίζω και υποστηρίζω την πρόταση του κυρίου Καράς να υπάρξει και χωρισμός, διαχωρισμός της ε, οδηγίας αυτής ένα τμήμα να αφορά την πολιτική αποδοχών και την ε, αντιμετώπιση των κινδύνων και αυτό μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2011 και χωριστά για τα υπόλοιπα θέματα. Και να είναι χωριστό το θέμα της ε, επανατιτροποίησης και της, των συναλλαγών συσχετισμού. Αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να καθυστερήσει και να το εξετάσουμε ενδελεχέστερα. Κάθριν Στάιλερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Συγήτρια. Ο κ. Σμιτ αναφέρθηκε σε παραμύθια. Μου φαίνεται σαν ιστορία τρόμου περισσότερο. Και δεν ξέρω αν θα έχει τέλος που θα λέει ζήσαν όλοι καλά και εμείς καλύτερα. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για τη δουλειά που έκανε και θέλει να έχουμε διαφάνεια και δικαιοσύνη. Και θέλουμε να εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά μέχρι τον Ιανουάριο του 2011. Αλλά έτσι που πάντα πράγματα, με την συνεδρία σε 9 Απριλίου και με τα τεκτενόμενα στη ΣΥΠΑ, πρέπει να καταλάβουμε για ποιο λόγο προτείνονται καθυστερήσεις. Και πολύ συχνά στην Επιτροπή μας έχουμε εκπροσώπους της Επιτροπής της Βασιλείας που δίνουν στοιχεία. Ίσως η Γραμματεία μπορεί να μας πει πότε θα ξανάρθει η Επιτροπή Βασιλείας στην Επιτροπή μας να δώσει κάποια στοιχεία. Θα ήταν κάτι πολύ χρήσιμο. Όσον αφορά την ψηφοφορία τη επόμενη εβδομάδα εφόσον είχαμε καθυστέρηση την περασμένη εβδομάδα, διότι τα καταφέραμε ελάχιστη να πάμε στο Στρασβούργο, λόγω του ηφαιστιακού προβλήματο, ίσω μια καθυστέρηση στην ψηφοφορία την επόμενη εβδομάδα να ήταν χρήσιμη. Α αποφασίσει η συγγήτρια όμως και ο Σκιώδης. Είναι ένα θέμα που αφορά του πολίτε μα και είναι κρισίμου σημασία στο να περάσουμε ένα ψήφισμα και αναμφισβήτητα οι κεφαλουχικές απαιτήσει που αισθάνονται πιστεύω ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι κεφαλουχικές απαιτήσει για να μην επαναληφθούν τα σφάλματα του παρελθόντος. Ευχαριστώ πολύ. Καλή τύχη ε, στην εισηγήτρια Γκούναρ Χόκμαρ. Ευχαριστώ. Θεωρώ καμιά φορά ότι όταν συζητάμε τη χρηματοδοτική αγορά, τις αγορές, τις θεωρούμε σαν να είναι απομονωμένες. Είτε κερδίζουν, είτε βλάπτουν την υπόλοιπη οικονομία. Έτσι το βλέπουμε και δεν ίσχυε αυτό. Ο κ. Σμιτ το ανέφερε και ο κ. Μπάρς αναφέρθηκε σε άλλη διάσταση. Τη, τη διατλαντική σχέση και πόσο σημαντική είναι. Πρόσφατα ελήφθη μια απόφαση που άλλαξε τους κανόνες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με ισχυρότερη θέση για την Κίνα και άλλες οικονομίες. Αυτό είναι μήνυμα αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στην οικονομία. Όταν συζητούμε αυτό το θέμα ή το επόμενο θέμα για τις κεφαλουχικές απαιτήσει και Βασιλεία 2, πρέπει να συζητήσουμε και τι συνέπειες που έχουν αυτά επί της οικονομίας εν γέννη, στο σύνολό της. Είχαμε τεράστια ε, χρηματοστική κρίση στην ευρωπαϊκή οικονομία. Ε, κανείς δεν ήταν ικανοποιημένος γι' αυτό πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα έχουμε νέα τέτοια κρίση. Διότι αν συμβεί κάτι τέτοιο εκ νέου θα δούμε ότι οι συνέπειες από το χρηματοπιστωτικό τομέα ε, μια νέα κρίση θα οδηγήσει νέα χρηματοπιστωτική αστάθεια. Αν έχει στέρηση η οικονομία μας ή αν μειωθεί η αξία των στοιχείων ενεργητικού, θα δημιουργήσουμε προβλήματα όχι μόνο στην πραγματική οικονομία μπορεί να διαχωριστεί από την χρηματοστική οικονομία αλλά και η χρηματοστική οικονομία. Και στέλνω μήνυμα στην εισηγήτρια και του σκιώδεις εισηγητέ που θα συναντηθούν να συζητήσουν τι τροπολογίε. Όλε αυτέ τι πτυχέ να τι λάβουν υπόψη. Τώρα συζητάμε στο Κοινοβούλιο το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 που απαιτούνται καινοτομίες, επενδύσεις και δεν θα πρέπει να τα λησμονούμε αυτά όταν θα συζητούμε και το ποσοστό της, της του φαινομένου μόχλευσης κλπ. Και, και τις τράπεζες. Διότι αν είμαστε υπερβολικά επιτυχείς ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους στο χρηματοστικό τομέα, θα πετύχουμε τη δημιουργία τεραστίων κινδύνων όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική ισορροπία και όσον αφορά την κοινωνία μας. Άρα οι συγγήτρια και οι συγγητέ, οι σκιώδει, α συζητήσουν τι τροπολογίε, λαμβάνοντα υπόψη το σύνολο τη οικονομία. Όχι μόνο τι χρηματοπιστωτικέ αγορέ. Ευχαριστώ. Wolf Klintz. Ähm, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να πω κάτι πάρα πολύ σύντομα. Ήμουνα το πρωί σε μια συνδιάσκεψη για τα χρήματα οικονομικά θέματα και φαίνεται ότι υπήρξε μια άποψη η οποία διατυπώθηκε και αποκρισταλώθηκε εκεί για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους για τις τράπεζες και αυτό φυσικά αναφέρεται και στην ε, οδηγία για την κεφαλουχική επάρκεια. Αν καταφέρουμε να οργανώσουμε έτσι τις τράπεζες ώστε όταν γίνεται κάποιο ατύχημα μέσα σε εισαγωγικά δεν θα πάρει μαζί του στην άβυσο όλο το πιστοτικό σύστημα να μπορέσουμε δηλαδή να αποσπάσουμε τα τμήματα τα οποία έχουν προβλήματα και το υπόλοιπο τμήμα της τράπεζας να μπορεί να λειτουργήσει. Τότε μπορούμε με μια αρκετά ε, σαφή και διάφανη διαδικασία να λειτουργήσουμε. Αυτό μου είπανε πολλοί ότι αυτό δεν γίνεται. Όταν ε, ε, μια τράπεζα πτωχεύει, πτωχεύει τελείως. όταν έχει προβλήματα με το τωρινό σύστημα δεν μπορεί να υπάρξει απόσπαση του κομματιού το οποίο μπορεί να έχει προβλήματα. Και επομένως ε, αστοχή σε αυτή την περίπτωση οποιαδήποτε εποπτεία τη τράπεζα. Αλλά μου φάνηκε μια ενδιαφέρουσα πρόταση να μπορούμε να αποσπούμε τμήματα από τι τράπεζε οι οποίε έχουν προβλήματα. Ευχαριστώ, λέει και πρόεδρο. Εγώ. Συνοψίσω τα σχόλιά μου, σα και Όδης του Άλντε και να συνοψίσω και τα ερωτήματα που ετέθησαν στη γραμματεία. Τα περισσότερα καλύφθηκαν. Ευχαριστώ την εισηγήτρια, διότι με ανοιχτό τρόπο βοήθησε τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων με τους σκιώδες. Ανοίγεται ένας δρόμος προς κοινή προσέγγιση, παρόλο που δεν έχουμε την ακριβή διατύπωση που θέλουμε σε κάθε σημείο. Απατώντας σε αυτό που είπε ο Γκούναρ Χόκμαρκ. Υπενθυμίζω στην Επιτροπή ότι στις ακροάσεις υπέγραψαν και ο Λιβρέν και ο Μισελ Μπαρνίε, δύο επίτροποι, υπέγραψαν, υποσχέθηκαν ότι θα εξετάσουν τις συνέπειες της νομοθεσίας που θα ακολουθήσει την κρίση. Και δεν αναφερόταν μόνο στο συγκεκριμένο κομμάτι του CRD και δεν αφορά μόνο τις κεφαλικές απαιτήσει, αλλά και ο συσχετισμός αυτού με όλα τα άλλα στοιχεία. Και ο συνδυασμός μπορεί να έχει πολύ μεγάλες συνέπειες και συμφωνώ με αυτά που υπόθηκαν. Προσπαθούμε να διαφυλάξουμε μέσω κεφαλαίου της τράπεζας, ταυτόχρονα εφευρίσκουμε εξόδους κινδύνου για κάποια τμήματα προς διάσωση και έχουμε άλλα τμήματα προς χεροκοπία και κατάρρευση και δημιουργούμε και διάφορους πόρους διάσωσης. Όλα αυτά καλά και άγια, αλλά αν τα συναθρήσουμε, δημιουργούνται πολλά προβλήματα ενδεχομένω. έτσι πιστεύω, μακροοικονομικά. Διότι μιλάμε για τεράστια ποσά χρηματικά που αφαιρούνται από την υποστήριξη πραγματικής οικονομίας. Για κάθε λίρα που βάζει στο Ταμείο Διάσωσης, βγάζεις 10 λίρες από την πραγματική οικονομία. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζουμε. Αλλά πρέπει να κάνουμε και κάτι. Συμφωνώ, χρειάζεται σταδιακή εφαρμογή. Και ίσως με, τέτοια, με κάποια μέτρα grandfathering πατρογονικά, κυρίως για να δουλέψει αυτό το κομμάτι του CRD. Σε ένα πρώιμο στάδιο είναι σημαντικό να διαφυλάξουμε για δραστηριότητες χαρτοφυλακίου κάποια κεφάλαια. Μεγάλα κέρδη εκ νέου γίνονται εκεί, σε αυτό το τομέα, και για άλλα επίμαχα νομοθετήματα, τι λέμε, λέμε τι θα πει το κοινό αν δεν κάνουμε κάτι, τι θα πει ο λαός. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και εδώ. Βλέπουμε τι αμοιβέ καταβάλλονται, τι πόνους καταβάλλονται. Είναι απαράδεκτο να μην κάνουμε κάτι όσον αφορά τα χαρτοφυλάκια συναλλαγών. Και η εναλλακτική όσον αφορά τα κεφάλαια είναι να γίνει ένας διαχωρισμός προς ξεχωριστές τράπεζες ε, επενδυτικές. Κάποιες χώρες συμφωνούν. Να πετύχουμε αυτό το διαχωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη θα είναι δύσκολο μάλλον. Άρα, θα πρέπει να δείξουμε στον κόσμο ότι είμαστε σοβαροί ότι θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτού του είδους ε, τραπεζικών δραστηριοτήτων τύπου καζίνο όπως αποκαλείται και Μιλάμε για επενδυτική τράπεζα, γιατί οι τράπεζες αυτές τι κάνουν, επενδύουν οι επενδυτικές τράπεζες. Επενδύουν και πετυχαίνουν αυτά που θέλουμε. Δεν θα πετύχουμε την υποδομή που χρειαζόμαστε για ενέργεια και για άλλους τομείς, αν δεν έχουμε αυτές τις τράπεζες που επενδύουν και κάνουν τη δουλειά τους. Αυτός μην το λησμονούμε. Πρέπει να κάνουμε κάτι και για τις αμοιβέ, για τα μπόνους, το ταχύτερο δυνατόν, όλοι συμφωνούμε. Και τέλος, μια προειδοποίηση. Ο κύριος Κάρας ήδη μας υπογράμμισε ότι έχουμε κάποιες εκκρεμότητες όσον αφορά την τιτλοποίηση. Και η γραμματεία τίμασε έναν κατάλογο όλων των εκκρεμών αναλύσεων που μας υποσχέθηκαν και που καθυστερούν και δεν λάβαμε κάποια εξήγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί δεν λάβαμε τις εκθέσεις και γιατί καθυστερούν. Γι' αυτό θα στείλω μία επιστολή, ίσως να εστάλει και σήμερα μία επιστολή και ζητώ εξηγήσεις. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι πολλές από τις ρήτρες αναθεώρησης είχαν μπει σε επίπεδο τριμερούς διαλόγου εν ώψη συμβιβασμού για να περάσει νομοθεσία. Άρα είναι σοβαρότατο ζήτημα αυτό. Θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε ρήτρε αναθεώρησης, ούτω ώστε να πετύχουμε συμβιβασμούς και συμφωνίες. Αν αμελούνται όλα αυτά τα σημεία ανεξήγητα. Εγώ το παίρνω πολύ στα σοβαρά. Το ότι αμελήθηκαν αυτές οι ρήτρες αναθεώρησης και δεν δόθηκε καμία εξήγηση. Γι' αυτό θα στείλω κι εγώ επιστολή. Προειδοποίηση είναι αυτή. Χρειαζόμαστε διαβεβαιώσεις σχετικά με εισαγόμενους μηχανισμούς για τη σταδιακή εφαρμογή των μέτρων. Αν έχουμε ρήτρες αναθεώρησης, ρήτρες ραντεβού κλπ. Αυτά έχω να πω. Και θα δώσω ξανά το λόγο στην Λίν, στην εισηγήτρια. Α, έχω κάποιες ε, ημερομηνίε να σας ανακοινώσω. Κάθριν, ο Γενικός Γραμματέας της Επιτροπής της Βασιλείας, στις 3 Μαΐου θα είναι σε ακρόαση για το CRD4 και το χρονοδιάγραμμα ποιος, θα το τίμαζε το χρονοδιάγραμμα που θα μπορούσαμε να έχουμε θα ήταν άλλη μια ανταλλαγή απόψεων στις 21 Ιουνίου και θα ακολουθήσει ψηφοφορία στην ΕΚΟΝ στις 22 Ιουνίου ή δυνατόν και ίσως στην Ολομέλεια του Ιουλίου την 1η του Σεπτεμβρίου. Αυτό είναι για να πάρετε μια ιδέα του χρονοδιαγράμματος που θα προταθεί. Α, τότε καλά. Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από τους συμβιβασμούς που θα πετύχουμε και τις συνεννοήσεις μεταξύ σκιωδών, μεταξύ των ομάδων δηλαδή. Θα τις κάνουμε όσο το δυνατόν συντομότερα. Εγώ θα προτιμούσα να ψηφίσουμε τον Ιούλιο για να έχουμε έτσι έξι μήνες μέχρι τα πράγματα να εγκριθούν. αλλά παρόλα αυτά σας είπα εξαρτάται. Και θα ήθελα τώρα να κάνω μερικά σχόλια στα δικά σας. Ακούστηκαν πολλά για την ανάγκη διεθνούς συνεργασίας. Ναι, φυσικά υπάρχει αυτή η ανάγκη αφού μιλάμε για ε, παγκόσμια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και δεν θέλουμε ή τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά να ζημιωθούν από τον διεθνή ανταγωνισμό. Αλλά δεν πρέπει να γνωρούμε ότι πολλές από τις εθνικές μας τράπεζες δεν έχουν επαρκή κεφάλαια. Εγώ δεν μιλάω υπέρ του τραπεζικού συστήματος, αλλά υπέρ ολόκληρης της οικονομίας. Χρειάζονται μεν τράπεζες που να λειτουργούν σωστά, αλλά όχι να τα βασίζουμε όλα να τα προσαρμόζουμε στις ανάγκες των τραπεζών. Ακόμη περιμένω να μου δώσουν οι τράπεζες τα στοιχεία που επανειλημμένως ζήτησα. Γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της προτινόμενης οδηγίας εγκαίρως. Δεν το κατάλαβα ακόμη. Νομίζω ότι και οι τράπεζες έχουν την υποχρέωση να μας δηλώσουν γιατί έχουν τα προβλήματα αυτά, γιατί δεν μπορούν να δανειοδοτήσουν ή αν έχουν επαρκή κεφάλαια. Είχαν ήδη 12 μήνες από τη Βασιλεία μέχρι τώρα και δεν μας απαντάνε. Επομένως δεν καθυστερούμε εμείς, αλλά δεν μπορεί να είναι συνεχής δικαιολογία ότι δεν απαντάνε οι τράπεζες. Νομίζω λοιπόν ότι θα καθορίσουμε από την 1η Ιανουαρίου 11 τους κανόνες και μετά θα δούμε πώς ακριβώς θα εφαρμοστούν. Ίσως προοδευτικά με phasing in. Αλλά έτσι θα είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρξει μία αύξηση του κεφαλαίου των τραπεζών και μετά βλέπουμε. Θα βρεθεί ένας μηχανισμός που να μην χρειάζεται καθυστέρηση. Εγώ δεν δέχομαι την καθυστέρηση. Θα συζητήσουμε τρόπους εφαρμογής όπως προοδευτική εφαρμογή, αλλά υπάρχουν δύο τράπεζες κύριε Σμιτ, δύο που πιέζουν ιδιαίτερα και λένε ότι πρέπει πρώτα να αυξήσουν το κεφάλαιό τους κατά 7 ή 10. Αν όμως χρειάζονται 700 ή 1000% παραπάνω κεφάλαιο, αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν επαρκή κεφάλαια ήδη. Και δεν το λένε. Εδώ δώσαμε εκατομμύρια για να βοηθήσουμε τις τράπεζες και στην έκθεσή μας εδώ λέμε απλώς ότι αν οι τράπεζες θέλουν να αναλάβουν περισσότερους ή μεγαλύτερους κινδύνους, τουλάχιστον να είναι βέβαιες ότι είναι σε θέση να πληρώσουν και σε περίπτωση προβλήματος. Και γι' αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα επιμείνουμε επί των αρχών τουλάχιστον της έκθεσης, ενώ θα είμαστε ελαστικοί στον τρόπο εφαρμογής. Και εγώ δεν θέλω να πτωχεύσουν οι τράπεζες, αλλά αν μόνο δύο από τις μεγαλύτερες βέβαια έχουν δημιουργήσει τα προβλήματα, δεν σημαίνει ότι θα τους δώσουμε και πλήρη δικαιώματα να κάνουν ό,τι θέλουν. Φυσικά δεν θέλουμε και άλλη κρίση, αλλά πρέπει να δούμε τα στοιχεία που δεν μας τα έχουν δώσει συχνά στις συζητήσεις και συναντήσεις που έχω με προσώπους τραπεζών μου λένε δεν μπορώ να σας δώσω αυτά τα στοιχεία γιατί είναι εμπιστευτικά και αν μας υποχρεώσετε να αυξήσουμε το κεφάλαιό μας δεν θα μπορέσουμε να δανειοδοτούμε ε, με τρόπο χρήσιμο. Και άλλοι μου λένε είναι θέμα δικής μας ευθύνης αλλά και εγώ έχω ευθύνη για τους εκλογείς μου και δεν θέλω τελικά όλα να τα πληρώνει ο φορολογούμενος. Υπάρχει λογική λύση. Και ο αρμόδιος επίτροπος είδε το σχέδιο έκθεσής μου και συμφωνεί. Ο συμβιβασμός που μπορεί να επιτευχθεί δεν είναι ότι θα υπάρξει απεριόριστη καθυστέρηση μέχρι όλες οι τράπεζες να μην έχουν πρόβλημα γιατί τελικά και αυτό θα το πληρώσει ως νύφη ο φορολογούμενος. Πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι και ρεαλιστές. με τις συζητήσεις που, είχα, από τις συζητήσεις που είχαμε τους Κιώδης κατάλαβα ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε λογικό συμβιβασμό που να καλύπτει όλα όσα είπαν οι συνάδελφοι σήμερα. Δεν θέλω όμως να διχτούμε πολύ μαλακοί γιατί έχουμε δει ότι όταν οι κανόνες λειτουργίας των τραπεζών είναι υπερβολικά ελαστικοί καταλήγουμε τελικά να δαπανούνται τα χρήματα του φορολογουμένου για να κάνουν οι τράπεζες την πίεση, το lobbying τους. Αυτά είναι απαράδεκτα. Δεν πρέπει να πληρώνει πάντα την ύφη ο φορολογουμένος. Μάλιστα ευχαριστώ. Το προτινόμενο χρονοδιάγραμμα που μπορεί βέβαια να αλλάξει είναι ότι Επιμένουμε στην κεφαλαιακή επάρκεια και η οδηγία για το CRD4 και την, και την επόμενη ανταλλαγή απόψεων θα την κάνουμε με εισηγητή τον κύριο Ότμαρ Καράς. Όχι, όχι θέλω να επανέλθω στον χρόνο, να επανέλθω. Διότι αν πάμε μέχρι το Σεπτέμβριο μετά, ιδιαίτερα για την απόδοση που όλοι συμφωνήσαμε ότι είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό και λεπτό και ευαίσθητο θέμα, είναι υπερβολή ο Σεπτέμβριος. Αν δεν μπορούμε να ψηφίσουμε πριν το Σεπτέμβριο, τότε είναι πολύ αργά. Είναι πολύ αργά. Και γι' αυτό νομίζω ότι το, χρονοδιάγραμμα που πρότεινε η Αιλίν είναι το σωστότερο. Μα θα προσπαθήσουμε για Ιούλιο. Αλλά τα πράγματα δεν γίνονται μεμονωμένα υπάρχουν και άλλες επιτροπές που πρέπει να γνωμοδοτήσουν και μπορεί να μην προλάβουν. Θα προσπαθήσουμε πάντως για Ιούλιο, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ό, μέχρι το CRD4, ο κύριος Καράς. Κυρία Πρόεδρε, ναι. Νομίζω ότι ήδη μας δείχνει πολλά η προηγούμενη συζήτηση. Είναι πολλά θέματα για τα οποία θα πρέπει να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει όλοι μαζί ομού να αντλήσουμε τα σωστά συμπεράσματα από την κρίση και με νυφάλιο τρόπο να εφαρμόσουμε τις κατάλληλες ρυθμίσεις. Και αυτό χρειάζεται λιγότερο συναισθηματική αντιμετώπιση. Είναι βέβαια είναι μια κατάσταση η οποία έχει δημιουργήσει πολλές ανησυχίες και πολλά συναισθήματα, αλλά εμείς πρέπει με αντικειμενικό και νυφάλιο τρόπο να τα αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά. Λοιπόν, έχουμε τονίσει ότι πρέπει το ταχύτερο δυνατό να βρούμε μια λύση για τα θέματα για, την, ε, για τις αμοιβέ των στελεχών, την πολιτική αποδοχών και πρέπει να μπορέσουμε να λύσουμε τα υπόλοιπα προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εφαρμογή των αποφάσεων. Δεν είπε κανείς ότι δεν θέλουμε να έχουμε μία απόφαση την 1η Ιανουαρίου 2011, μία απόφαση για την πολιτική αποδοχών. Τονίσαμε στην τελευταία μας συνεδρίαση πόσο σημαντικό είναι να μπορέσουμε να πάρουμε μία πρωτοβουλία για τα θέματα αυτά και να μπορέσουμε να συζητήσουμε σε συνεκτικό επίπεδο τα θέματα αυτά. Τώρα έχουμε τη συζήτηση για το CRD3, για την οδηγία για την κεφαλογική επάρκεια. Έχουμε τώρα την ε, ΣΥΑΔΙ 4 και την Επιτροπή της Βασιλείας που είναι το επόμενο θέμα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητάει παράλληλα θέματα τα οποία δεν πιστεύω ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μια πραγματική νομοθετική πρόταση όμως η οποία θα μας επιτρέψει να επηρεάσουμε την πολιτική. Ο στόχος της δικής μας εκθέσεως πρωτοβουλίας που δεν είναι νομοθετική ακόμα είναι παράλληλα με, την, παράλληλα με τη συζήτηση για το CRD3 αλλά και παράλληλα με αυτά τα οποία κάνει η Επιτροπή της Βασιλείας να παρουσιάσουμε τις δικές μας πρωτοβουλίες ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί με τον τρόπο αυτό μπορούμε να δείξουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ενεργά εμπλεκόμενο στην συζήτηση αυτή και θέλουμε να ασκήσουμε επιρροή και όχι απλώς να αντιδρούμε και να εφαρμόσουμε τις αποφάσεις, τις αποφάσεις των άλλων. Μπορούμε λοιπόν αυτή την έκθεση να τη χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα για πολιτική διευκρίνηση της πορείας που θέλουμε να ακολουθήσουμε στην νομοθετική διαδικασία όπου θα εμπλακούμε πλήρως ως Κοινοβούλιο. Αυτός νομίζω πρέπει να είναι ο στόχος μας να υπάρξει ένα συντονισμό μεταξύ Κομισιών, Επιτροπής Βασιλείας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό θα ενισχύσει και την Κομισιόν μέσα στο ρόλο της ε, συντονιστικής της εργασίας στα πλαίσια της Επιτροπής Βασιλείας και φυσικά θα αυξήσει και την επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην, Βασιλεία. στην Επιτροπή της Βασιλείας. Το είδαμε αυτό στο επίπεδο της Βασιλείας 2. Είχαμε πραγματικά ένα σημαντικό ρόλο ως Ευρωπαϊκή Ένωση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εξασφαλίσαμε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο χάρη και στη συζήτηση η οποία έλαβε χώρο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για να γίνουν λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να υπάρξει ένα σωστό σχεδιασμό των μεμονωμένων προτάσεων και θα πρέπει να τονίσουμε ότι η αποφάση των G20 για την ποιότητα του κεφαλαίου και τη ρευστότητα θα πρέπει να εφαρμοστούν όπως και τα αντικυκλικά ε, μέτρα για τράπεζες που έχουν μεγάλη σημασία συστημικά και οι οποίες παραμένουν ακόμα να καθοριστούν ποιε είναι. Τώρα για το CRD3, για το CRD3 αυτός είναι ένας τομέας όπου θα πρέπει να υπάρξει και έκθεση αντικτύπου και θα πρέπει να υπάρξει και μια μελέτη <clears throat> αντικτύπου η οποία δεν θα περιορίζεται μονάχα στον τραπεζικό τομέα αλλά θα περιλαμβάνει και τις επιπτώσεις τις ευρύτερες για την πραγματική οικονομία. <clears throat> Μετά από την κρίση δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία ότι θα πρέπει να επανεξεταστούν οι προδιαγραφές της Βασιλείας 2 και να αντλήσουμε τα απαραίτητα συμπεράσματα από την κρίση. Θα πρέπει να εξεύγουμε την κατάλληλη ισορροπία. Είναι σαφές ότι είναι απαραίτητα τα μέτρα αυτά, αλλά είναι απαραίτητο να συνδυάσουμε αυτές τις αποφάσεις με άλλες νομοθετικές αποφάσεις αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι η ανάπτυξη στην πραγματική οικονομία και η ικανότητα των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη της οικονομίας και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξουν και συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών για τα θέματα αυτά. Τονίζω λοιπόν ότι αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας είναι ένα πολιτικό κομμάτι αυτής της ε, σειράς προτάσεών μας και είναι μια ευκαιρία να μπορέσουμε να διευκρινίσουμε ορισμένα θέματα ουσίας. Θέλουμε να έχουμε ένα νέο ορισμό για το τι ακριβώς πρέπει να είναι το κεφάλαιο το οποίο υπόκειται σε κεφαλογικές ε, ε, απαιτήσει και πρέπει να έχουμε και ένα χρονοδιάγραμμα για όλα αυτά τα θέματα. Θα πρέπει πάντα να περιλαμβάνεται και η πτυχή του κινδύνου όταν συζητάμε για κεφάλαιο. Αυτό είναι μία, ένα από τα διδάγματα της ε, κρίσης. Η κρίση ήταν και μια κρίση ρευστότητος και όχι μια κρίση κεφαλαιοηχική επάρκειας. Και εδώ πρέπει να εξασφαλίσουμε και μια ισορροπία μεταξύ επάρκειας κεφαλαίου και ε, ρευστότητος. Το να έχουμε απλώς ένα ε, ποσοστό μόχλευσης χωρί εκτίμηση των κινδύνων και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και επίση θα πρέπει να αποφύγουμε να παίρνουμε μέτρα τα οποία σε μια κρίση θα δράσουν υπερκυκλικά. Είναι απαραίτητο λοιπόν να κάνουμε και μια διάκριση μεταξύ διαφορετικών τραπεζών. Δεν μπορούμε να έχουμε μια συλλήβδη πολιτική one size fits all που να καλύπτει όλες τις τράπεζες. Έχουμε διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία έχουν βοηθήσει την εξασφάλιση της ισορροπίας στην Ευρώπη μέσα στην οικονομική κρίση και πρέπει να τα λάβουμε αυτά υπόψη. Και πρέπει επίση να δούμε και ποια είναι η διάδραση μεταξύ των προτάσεων για τη ρευστότητα και των απαιτήσεων κεφαλαίου. Όλα αυτά θα πρέπει να τα ερευνήσουμε. Επίση, μπορούν να είναι χρήσιμε μεταβατικέ ρυθμίσεις για να μπορέσουν να βοηθήσουν τι τράπεζε, να περάσουν στι νέε ρυθμίσει και να αποκτήσουν το κατάλληλο κεφαλαίο. Όπω είπε και ο Βολφ Κλίντς, υπήρξε αυτό το εργαστήριο που διοργάνωσε η Κομισιόν και η Κομισιόν έκανε μια διαδικασία διαβούλευσης στην οποία έλαβε 135 απαντήσεις από διάφορους φορείς και αυτό θα ήταν χρήσιμο να το εξετάσουμε. Θα πρέπει να ξέρουμε λοιπόν ποια είναι τα βασικά θέματα. Πρότυπα για τη ρευστότητα, ορισμός του τι αποτελεί ίδιο κεφάλαιο, ε, ποσοστά μόχλευσης, ο κίνδυνος, ε, πιστοτικός κίνδυνος αντισυμβαλωμένου, αντικυκλικά μέτρα, τα πιστοτικά ιδρύματα τα οποία έχουν μεγάλη σημασία για το σύστημα και το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις τράπεζες. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας για να μπορέσουμε να θέσουμε τις πολιτικές μας προτεραιότητες, για να καθορίσουμε τις απαραίτητες έννοιες οι οποίες είναι οι σωστές, ώστε να βοηθήσουμε την Κομισιόν και την Επιτροπή Βασιλείας και τις χώρες μέλη μας για να λειτουργήσουν σωστά στη διαδικασία της Βασιλείας και αυτό νομίζω θα είναι ένα από τα σημαντικότερα στάδια εν ώψη της νομοθετικής πρότασης που θα έρθει από την Κομισιόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και φυσικά με την έκθεσή μας θέλουμε να βοηθήσουμε και την Κομισιόν να ενισχύσει τη θέση της. Πώς πάει το χρονοδιάγραμμα τώρα. Η πρώτη συζήτηση γίνεται σήμερα, 26 Απριλίου, αναφέρθηκε στη συνέχεια 3 Μαΐου, να υπάρξει στη συνέχεια μία ακρόαση με εκπροσώπους του τραπεζικού τομέα, εκπρόσωπο του ΟΣΑ, εκπρόσωπο της Επιτροπής της Βασιλείας και άλλους εκπροσώπους σε αυτήν την ε, ακρόαση. Η... Το σχέδιο έκθεση θα πρέπει να είναι έτοιμο τέλη Μαΐου αρχές Ιουνίου. Η προθεσμία για τις τροπολογίες 28 Μαΐου 21-22 Ιουνίου θα γίνει η εξέταση των τροπολογιών, ώστε να μπορέσουμε να κλείσουμε το θέμα της CRD3, της Οδηγίας Κεφαλογικής Επάρκειας και να μπορεί να υπάρξει απόφαση στην Επιτροπή μας το Σεπτέμβριο και να πάμε στην Ολομέλεια τον Οκτώβριο. Αυτό είναι το τωρινό χρονοδιάγραμμα. Δεν προσπαθούμε να κάνουμε αγώνα δρόμου, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε σαφή την άποψή μας για τους πολιτικούς στόχους αυτού του, αυτής της ρύθμισης, ώστε να έχουμε μια ανοιχτή, διάφανη και συνεκτική ρύθμιση στον τομέα αυτό. Αυτό είναι ακριβώς ο στόχος της έκθεσης πρωτοβουλίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στους κοιόδης τώρα. Ούντο Μπούλμαν. Εξαφανίστηκε. Πού είναι Ούντο. κύριος Μπάλτ είναι ο επόμενο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Για το CRD3 έχουμε συζητήσει, συζητάμε τώρα, για το 4 δεν έχουμε ακόμα καμιά συγκεκριμένη πρόταση από την Κομισιόν. Νομίζω ότι η Κομισιόν όμως δεν ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση. Το να υπάρχουν συγχρόνως πιο αυστηροί ορισμοί για το ίδιο κεφάλαιο. Και από την άλλη μεριά, το να έχουμε ε, περιορισμούς, να έχουμε αύξηση του, των ε, κεφαλαιοχικών επαρχιών, το επίπεδο αυτού μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα. Δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να εκτιμούμε στο μέλλον έτσι την ανεξάρτητα το επίπεδο κεφαλοχικής επάρκειας. Όλα αυτά μπορούν να κινδυνεύσουν να οδηγήσουν σε ε, ανταγωνισμό, σε αθέμητο ανταγωνισμό μεταξύ πιστοτικών ιδρυμάτων που έχουν διαφορετική νομική μορφή. Λοιπόν, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις διαφορές αυτών των ιδρυμάτων και επίσης δεν έχουμε ακόμα τις λεπτομέρειες της ε, πρότασης της Κομισιόν και νομίζω ότι η εισαγωγή ενός ορίου στο στο επίπεδο μόχλευσης, αυτό είναι μια πολύ κακή ιδέα. Αυτό είναι αντίθετο με αυτά τα οποία αναφέρει και η Βασιλεία 2. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε παράλληλα και ποσοστό μόχλευσης και αιτήσει κεφαλαιοχικής επάρκειας. Αυτό μπορεί σε ορισμένε περιπτώσεις να οδηγήσει σε, σε ανάληψη μεγαλύτερων κινδύνων από ορισμένου. Και τέλος, σε σχέση με την αβεβαιότητα που υπάρχει σε σχέση με την εφαρμογή του CRD3 θα πρέπει να μην το υπερφορτώσουμε αυτή τη στιγμή υπερβολικά το, τη ρύθμιση και τα θέματα αυτά. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς έχουν εφαρμοστεί μέχρι στιγμή τα διάφορα νομοθετήματα, που είναι τα κενά τα οποία έχουν και πώς έχει αντιδράσει η αγορά στα θέματα αυτά. Χρειάζεται λοιπόν μια συνολική αποτίμηση και πιστεύω ότι μόνο επί τη βάση μιας συνολικής έκθεσης αντικτύπου θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε για το θέμα αυτό και γι' αυτό υποστηρίζω πλήρως αυτά που είπε ο Όθμαρ Καράς. Προσπαθώ να δω αν έχουμε σκιώδεις που ζητούν το λόγο. Όχι. Α, η Βίκη. Ευχαριστώ. Πάλι αυτά τα θέματα CRD3, CRD4 και κατά πόσο θα πρέπει να εφαρμοστούν διεθνώς πρότυπα και θα πρέπει να δούμε και τις ορευτικές συνέπειες των διαφόρων επιπέδων μεγεθών κεφαλαίων που διατίθεται στις τράπεζες. Τώρα τα έγγραφα διαβούλευσης και το έγγραφο εργασία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή του CRD4. Είναι σημαντικά κάποια στοιχεία που ταιριάζουν με αυτό που συζητάμε, ο ορισμός του, του ποσοστού μόχλευση, κίνδυνο ε, των ε, συμβαλωμένων μερών, αντικυκλικό κεφάλαιο, συστημικές τράπεζες κλπ. Τα έχουμε κουβεντιάσει. Και στο θέμα EBA και στο ψήφισμα και, τον ενίο, και τους κανόνες. Ε, αυτή δεν είναι απομονωμένη η νομοθεσία, ταιριάζει και με άλλες πτυχές. Και στη Βασιλεία θα εξετάσουν τον αντίκτυπο. Τώρα όσον αφορά τη ρευστότητα. Η κρίση, η χρηματοστατική κρίση ξεκίνησε σαν κρίση ε, ε, πιστοτική, αλλά γρήγορα έγινε κρίση ρευστότητα, γιατί στέγνωσαν οι αγορέ. Τα χρηματοστικά ιδρύματα μάθαμε ότι θα πρέπει να έχουν ρευστό. Άρα τι είδους ε, ρευστά στοιχεία ενεργητικού πρέπει να έχουν. Και έχουμε ένα φαύλο κύκλο μπροστά μας για την ώρα. Όσο πιο πολύ κρατούν χρέος κυβερνητικό οι τράπεζες, δημιουργείται ζήτηση για κυβερνητικό, για κρατικό χρέος. Και πολλές κυβερνήσεις αυξάνουν το κρατικό χρέος, όπως και στη δική μου χώρα. Άρα γίνεται ένας ε, φαύλος κύκλος εντός των χρηματοστηρικών αγορών. Η ρευστότητα λοιπόν και η ανάγκη ενός γενικού ποσοστού μόχλευσης. Τα στοιχεία ενεργητικού με σταθμισμένο κεφάλαια του CRD δεν έλαβαν υπόψη τη, γενικό, τη γενική μόχλευση, διότι μπορεί να είχαν χαμηλή στάθμιση, όπως χρέη στεγαστικών δανείων, που είχαν άλλα επίπεδα μόχλευσης και ίσως να είχαμε υποτιμήσει ε, το κίνδυνο στις κεφαλοχικές απαιτήσει. Ε, χρειάζεται ένας γενικός έλεγχος μόχλευσης. Θα ήταν λογικό κάτι τέτοιο. Πρέπει να καταλάβουμε όμως ότι κάποιοι κίνδυνοι είναι λιγότεροι κίνδυνοι από άλλους κινδύνους. Άρα κάποιοι κίνδυνοι ίσως να είναι πιο αποδεκτοί. Αν αγοράζει κανείς ένα σπίτι, παραδείγματος χάρη, μπορεί να πάρει περισσότερο χρέος και λιγότερο ρευστό από ό,τι για να πάρει ένα αυτοκίνητο. Διαφορετική αντιμετώπιση. Επειδή ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές των ακινήτων, ε, είναι μικρότερο ο κίνδυνο για το στοιχείο ανεργητικού από ό,τι ένα αυτοκίνητο. Μόχλευση και ρευστότητα λοιπόν που εξεταστούν. Και άλλα θέματα, αυτή η γενική ανησυχία που επικρατεί, ότι δεν έχουμε γενικά πρότυπα, παγκόσμια πρότυπα λογιστικών υπολογισμών. Άρα αυτό που λέει μια χώρα στις τράπεζες μπορεί να ερμηνεύεται διαφορετικά σε άλλη χώρα, διότι υπάρχουν διαφορετικά λογιστικά συστήματα. Ορισμός του κεφαλαίου πρέπει να εξεταστεί. Και με προτεραιότητα του CRD3 ζητάμε στις τράπεζες να αυξήσουν το κεφάλαιο. Αλλά δεν είναι ξεκάθαρο τι είναι αυτό το κεφάλαιο, ποιος είναι ο ορισμός του κεφάλαιου, ποιος θα είναι στο μέλλον. Θα θεωρούσε κανείς ότι κεφάλαιο στα πλαίσια του CRD3 θα εκάλυπτε απώλειες σε μία ύφεση. Όμως, το κεφάλαιο επίπεδου 2 δεν οδηγούσε σε απώλεια αυτούς που είχαν αυτό το από τη στιγμή που η τράπεζα ε, συνέχιζε δραστηριότητε. Τα χρήματα του φορολογουμένου πάνε στις τράπεζες για να τις βοηθήσουν και εκείνοι που έπρεπε να υποστούν τις συνέπειε και τις απώλειε τελικά δεν υπέστησαν καμία απώλεια. Άρα πρέπει να δούμε ποιο είναι ο θεμελιώδης ορισμός του κεφαλαίου. Διαφορετικά υπάρχει αβεβαιότητα στις τράπεζες. Δηλαδή τι κεφάλαιο προσπαθούν να συσσωρεύσουν. Και αυτή η αβεβαιότητα δεν τις βοηθά για δυνα... αντικυκλικό κεφάλαιο και δυναμικό εφοδιασμό. Είναι λογικό να δημιουργηθούν αποθέματα, αποθεματικά, εγκαίρως, ούτως ώστε όταν πάνε δύσκολα τα πράγματα να απαλύνονται οι απώλειες. Και εδώ παίζουν ρόλο και οι λογιστικοί κανόνες εγώ δάνειζα χρήματα και ανησυχώ γι' αυτό. Ίσως δημιουργήσουμε ένα μοντέλο που οδηγεί σε μεγαλύτερη δανειοδότηση. Αν μέσω ιστορικών απολειών προσπαθεί να προβλέψεις μελλοντικέ απώλειες ίσως να σπρώχνεις κεφάλαια, ε, να προωθεί χρήματα και δημιουργείς φυσαλίδες και στο μέλλον. Ιστορικές ιστορικέ δεν είναι καλή βάση απαραίτητα για προβολές προς το μέλλον όσον αφορά τι απώλειες. Το έγγραφο αναφέρεται σε συστημικά σημαντικά χρηματοστικά ιδρύματα που παραπέμπει και στα έγγραφα για τη διέξοδο από την κρίση. Και ήταν δύσκολο να καθορίσουμε ποια είναι τα συστημικά σημαντικά χρηματοστικά ιδρύματα. Δεν πρέπει να έχουμε υπόψη μόνο τις τράπεζες, αλλά και άλλους χρηματοψητικούς θεσμούς, θεσμικά όργανα, φορείς, σημαντικούς παράγοντες της χρηματοστικής ε, αγοράς, που εκεί ίσως να δημιουργείται συστημικός κίνδυνος και για το κεφάλαιο των αντισυμβαλωμένων μερών. Έχουμε κεντρικούς φορείς συμψηφισμού και πρέπει να εξεταστεί αυτό το θέμα σαν προτεραιότητα. Υπάρχουν πραγματικές επιχειρήσεις που στην αγορά παραγόγων ε, θέλουν να ξέρουν πόσο κεφάλαιο πρέπει να συσσωρεύσουν έναντι αυτών. Συγγνώμη, αυτά είχα να πω. Καθυστερούμε πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Και αυτό με ανησυχεί. Γιατί είναι πολύ σημαντικά θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε βέβαια και γι' αυτό δεν σας διακόπτω. Αλλά θα έχουμε κρίση χρόνου κάποια στιγμή αργότερα. Σας παρακαλώ λοιπόν να είστε το δυνατόν συντομότεροι και γι' αυτό εγώ δεν θα λάβω καθόλου το λόγο. Μπορώ να πω ότι σύμφωνα με πολλά από αυτά τα οποία ελέγχθησαν ήδη, ιδίω για τα ιστορικά θέματα, ο Ούντο Μπούλμαν, σε σου καθώς το λόγο, αλλά έλειπες προηγουμένως. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα ακολουθήσω τη μετριοπάθεια σας και θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Εγώ είχα δύο πράγματα να πω στον εισηγητή. Καταρχήν, στο διαδικαστικό επίπεδο υποστηρίζουμε απόλυτα την ιδέα να εργαστούμε ήδη τώρα και όχι να ξεκινήσουμε τη δουλειά μας όταν μετά από διεθνείς ε, διασκέψεις που δεν έχουν έτσι και καμία δημοκρατική εντολή, όπως εμείς που είμαστε νομοθέτες, βγουν αποτελέσματα. Θέλουμε ήδη τώρα σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να πούμε τι θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο και γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε μια παράλληλη εργασία μαζί με την Επιτροπή, παράλληλα με την Επιτροπή της Βασιλείας. Σε επίπεδο περιεχομένου. Ναι, υπάρχουν δυσκολίες, το τόνισαν πολλοί συνάδελφοι υπάρχουν δυσκολίες για το πώς λειτουργεί η ευρωπαϊκή κεφαλαία αγορά, αντίθετα από την αμερικανική κεφαλαία αγορά και υπάρχουν φυσικά και δυσκολίες επειδή τα χρηματοπιστωτικά μας ιδρύματα έχουν διαφορετικές ε, παραδόσεις, λειτουργούν με διαφορετικούς μηχανισμούς στα κράτη μας μέλη, αλλά πιστεύω ότι δεν πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε παντού εξαιρέσει. Αν κάνουμε για το κάθε τι εξαιρέσει, κάνουμε ακριβώς αυτό το οποίο δεν θέλουμε. Αφήνουμε την Επιτροπή της Βασιλείας να πάρει τις αποφάσεις και να επιβάλλει ρυθμίσεις οι οποίες θα ισχύουν για τα χρηματοπιστωτικά μας ιδρύματα και αυτό δεν νομίζω ότι είναι το καλύτερο για μας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν λέμε ότι ο ορισμός του κεφαλαίου είναι ένα επίμαχο θέμα, βλέπουμε ότι στη Γερμανία υπάρχει πάντα ένα θέμα με, τις, ε, με τις, τα αποθεματικά τα οποία τίθενται σε επίπεδο κεφαλαίου. Βλέπουμε ότι στην περίπτωση της Βασιλείας υπάρχει κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με το νομικό, νομική ιδιότητα ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Αυτό δεν νομίζω ότι μας Μα διαφωτίζει ιδιαίτερα. Άμα κινδυνεύει να χρεοκοπήσει κάποιο ίδρυμα, πρέπει να το βοηθήσουμε. Επίση για τη μόχλευση. Εγώ θα υποστήριζα να λάβουμε υπόψη την ανάγκη να υπάρχει ένα μαξιλαράκι κατά κάποιο τρόπο από το τραπεζικό σύστημα, να παίξει ένα αντικυκλικό ρόλο το τραπεζικό σύστημα. Αυτό μας, δι... μας έδειξε η κρίση και θα σταματήσω εδώ για να μην ξεπεράσω το χρόνο μου.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 Μα γιατί μου ζητάτε να μιλήσω. Γιατί νόμισα ότι είδα το χέρι σας. Πρώτα σκιώδης είπαμε λοιπόν. Α, μάλιστα καλά. Α, τότε καλά. Πριν μιλήσω για την ουσία θα ήθελα να αναφερθώ στην παρουσίαση του Όθμαρ Καράς. Για μας τους πράσινους η έκθεση του είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τοποθετηθεί πριν λήξουν οι διαπραγματεύσεις στην Επιτροπή της Βασιλείας. Έχουμε λοιπόν επιτέλους την ευκαιρία να αποφανθούμε πριν αποφασιστούν τα πράγματα και άρα να πούμε και εμείς το λογάκι μας. Και πρέπει να επωφεληθούμε από αυτήν την έκθεση πρωτοβουλίας που είναι, είναι ιδιαίτερα καλό που ο εισηγητής είναι ο κύριος Καράς που έχει αξιοπιστία για να ακουστεί η φωνή του και προς τα έξω ως φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βέβαια. Αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας λοιπόν θα γίνει βέβαια αντικείμενο συμβιβασμού μεταξύ πολιτικών ομάδων αλλά έτσι θα αυξηθεί το, η σημασία της ε, προς τα έξω και θα αποτελέσει μοχλό για περισσότερη επιχειρηματολογία. Επί της ουσίας τώρα, για το περιεχόμενο δηλαδή, χωρίς να πω στις λεπτομέρειες, νομίζω ότι πρέπει, εκτός αν δεν κατάλαβα καλά το πλαίσιο που καθόρισε για την έκθεση του κύριου Καράς, Πρέπει φυσικά να αναφερθούν οι κύριες πολιτικές αρχές για τις κυκλικές συνέπειε και για τις μοχλεύσεις και αναμοχλεύσεις να υπάρξει κάποιος ορισμός του τι κεφάλαιο πρέπει να διαθέτει κάθε τράπεζα κτλ. Αλλά και επίσης πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε και ένα πιο τεχνικό ορισμό. Ω, βέβαια στην έκθεση αυτή πρωτοβουλίας δεν θα τα καλύψουμε όλα για το CRD4, και τις απαιτήσεις που έχουμε για κεφαλαιακή επάρκεια, αλλά ορισμένα σημεία της συμφωνίας τουλάχιστον που θα έχουμε πετύχει μεταξύ ομάδων να αναφερθούν για να επηρεάσουν αν μπορούν ή όσο μπορούν και τις διαπραγματεύσεις της Βασιλείας. Έτσι νομίζω ότι θα έχουμε προχωρήσει και αυξήσει την επιρροή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμείς βέβαια είμαστε υπέρ πολλών συμπερασμάτων των συζητήσεων στη Βασιλεία, όπως η θέληση να μειωθεί ο κυκλικός χαρακτήρας της πρότασης και η απέτηση αυτή της κεφαλαιακής επάρκειας συνδυασμό με την εκτίμηση του κινδύνου και επίσης είμαστε υπέρ μιας σφαιρικής μοχλεύσεως. Μπορεί βέβαια μερικοί αυτό να το θεωρούν περιττό διότι αν αυξηθεί το κεφάλαιο των τραπεζών δεν μπορεί να μην χρειάζεται αυτό που λέω. Αλλά εμείς νομίζουμε ότι χρειάζονται και τα δύο γιατί δεν ταυτίζονται. Εφόσον μάλιστα στην Ευρώπη δεν θα είναι εύκολο να απαντήσουμε τα θέματα της αντιμετώπισης των πιτοχεύσεων και δεν μπορούμε στην Ευρώπη να μεταφέρουμε ως έχει το αμερικανικό πρότυπο. Δεν ισχύει η αρχή το too big to fail. Δεν ισχύει. Και γι' αυτό πρέπει να μειωθεί ο, η έκθεση ορισμένων τραπεζών στους κινδύνους. Διάφορους κινδύνους. Είτε από την κεφαλαιακή επάρκεια είτε από άλλα μέσα. Υπάρχει λοιπόν έτσι εδώ πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Εμείς πάντως είμαστε υπέρ και των δύο τύπων νομοθέτησης και της μοχλεύσεως και του κεφαλαίου. Τέλος, θα προσέξουμε ιδιαίτερα ο ορισμός των κινδύνων που αφορούν το trading book να βασίζεται και σε μία ανάλυση της εμπειρίας που είχαμε μέχρι τώρα να υπάρξει δηλαδή μια επανεξισορρόπηση των κινδύνων όπως τους αποτιμούν οι τράπεζες και επ' αυτού θα επιμείνουμε ιδιαίτερα ως πράσινοι και πράσινες. Ευχαριστώ ο Γκούναρ Χόκμαρ, ευχαριστώ για την υπομονή σου. Ουδέν πρόβλημα, διότι μπορώ να εξοικονομήσω χρόνο λέγοντας συμφωνώ με τα περισσότερα από αυτά που υπόθηκαν και να προσθέσω κάποια πράγματα μπορώ να πω ότι θα ήθελα να υποστηρίξω τη στρατηγική της, ε, του εισηγητή όσον αφορά την αξιολόγηση συνεπειών, να εξεταστούν οι συνέπειες των συζητουμένων. Να προσθέσω κάποιες ε, πτυχές που πρέπει να σκεφτούμε. Σε αυτή την Επιτροπή συχνά μιλάμε για και υπογραμμίζουμε την ανάγκη για ευκολότερη ε, χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και πρέπει αυτό να το έχουμε υπόψη όταν μιλάμε για κεφαλουχικές απαιτήσει. Διότι δεν υποτίθεται κάνουμε το αντίθετο που ίσως να οδηγεί σε αντιφατικά αποτελέσματα. Αυτό θα έπλητε την πραγματική οικονομία και τη χρηματοπιστωτική οικονομία. Πρέπει λοιπόν να θυμόμαστε ότι υπάρχουν διαφόρων ειδών κινδύνοι. Και υπάρχει μια τάση και ένα κίνημα θα έλεγα να συζητούμε περισσότερο τα ποσοστά μόχλευσης και όχι την ανάλυση κινδύνου. Αυτό δεν θα βοηθήσει. Στις τελευταίες συζητήσεις ξεκινήσαμε λέγοντας ότι έχουν λίγα κεφάλαια οι ευρωπαϊκές τράπεζες. Είναι δύσκολο να λέμε κάτι τέτοιο. Αυτό συνεπάγεται ότι ξέρουμε ποια είναι η σωστή κεφαλουχική απέτηση. Και δεν είναι εύκολος αυτός ο καθορισμός, διότι εξαρτάται από τους κινδύνους που αναλαμβάνονται και εξαρτάται και από κάτι άλλο. Μπορούμε να λέμε ότι όσο πιο πολλά κεφάλαια έχουν οι τράπεζες, το καλύτερο. Μέσα σε μια στενή προπτική. Αλλά αυτό οδηγεί στο κίνδυνο ότι δίνουμε λίγα κεφάλαια στην οικονομία. Διότι χρειαζόμαστε κεφάλαιο στην αγορά για επενδύσεις, για καινοτομία. Η στρατηγική του 2020 υπογραμμίζει την ανάγκη να ηγηθούμε να χρηματοδοτήσουμε καινοτόμα προγράμματα. Όσο λιγότερα κεφάλαια έχουν οι όσο περισσότερα κεφάλαια έχουν οι τράπεζε, τόσο λιγότερα κεφάλαια θα έχουμε τι επενδύσει που απαιτούνται. Που είναι κρίσιμη σημασία για την οικονομική και χρηματοδοτιστική ισορροπία τη Ευρωπαϊκή οικονομίας. Να μην το λησμονούν αυτό. Διαφορετικά, στο τέλο, θα χάσουμε θέσει εργασία ανάπτυξη και οικονομική σταθερότητα. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η βασική απειλή όσον αφορά την χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι τα τεράστια ελλείμματα των δημοσιονομικών. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το είπε αυτές τις προάλλες. Όταν επικρατεί, κατάσταση επικρατεί σε κάποιες χώρες, δεν υπάρχουν κεφαλουχικές απαιτήσει επιτραπεζών που θα έλυναν το πρόβλημα της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Χρειάζεται σειρά δραστηριοτήτων για την επίτευξη του στόχου. Τέλος. Όταν συζητούμε τις συνέπειες των αυξημένων κεφαλοχικών απαιτήσεων πρέπει να ακολουθήσουμε ευρύτερη προσέγγιση. Μιλάμε τώρα για τράπεζες, θα μιλήσουμε για επιχειρήσεις ασφαλιστικές και θέματα φερεγγιότητας. Και εκεί θα συζητήσουμε το δύο θέμα των αυξημένων κεφαλουχικών απαιτήσεων. Οι ασφαλιστικές εταιρείες, ο τομέας αυτός, Εκεί υπήρξε πρόβλημα κεφαλουχικών απαιτήσεων, αλλά αυξάνονται κεφαλουχικές απαιτήσει. Η συνολική συνέπεια όλων αυτών μπορεί να μας οδηγήσει στην κατάσταση όπου οι πολιτικές αποφάσεις δίνουν λίγα ποσά στην οικονομία, λίγες επενδύσεις. Πρέπει να πετύχουμε τη σωστή ισορροπία. Γι' αυτό είναι σημαντικό που διεξάγεται η συζήτηση περί αναλύσεως αντιχτύπου. Χρειάζεται και ευρύτερη προσέγγιση. Δεν μπορούμε να θεσπίζουμε νοθεσία μόνο λαμβάνοντας υπόψη τι τράπεζε. Πρέπει να συζητούμε και να νομοθετούμε έχοντα υπόψη όλη την ε, εικόνα. Πώ μπορεί να ωφεληθεί από δυναμικέ και σταθερέ χρηματοπιστωτικέ ε, αγορέ η οικονομία. Ε, εσύ έχει το λόγο, Αλήν. Θα είμαι σύντομη λόγω χρονικών περιορισμών. Αλλά υποστηρίζω την προσέγγιση που ακολουθήθηκε τον κύριο Καρά, την ισορροπία μα. η εμπειρία μα από το CRD3 μα έδειξε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε έκθεση ίδια πρωτοβουλία ότι θα πρέπει να διεξάγονται ακροασει να γίνεται ανάλυση εξολογήσει ε, αντιχτύπου, διότι αυτό εξασφαλίζει το Κοινοβούλιο και αυτή η Επιτροπή ε, δίνει εντολή κατά κάποιο τρόπο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και βάσει της αναλύσεως αυτή, ούτω ώστε να δουν ποιο θα έπρεπε να είναι το περιεχόμενο και η προσέγγιση όσον αφορά το CRD3 πριν καταλήξουμε σε απόφαση τη ομάδα βασιλεία. Υποστηρίζω λοιπόν την προσέγγιση του εισηγητή και προφανώ θα την υποστηρίξουμε και σχετικά με τη σύνδεση που έχει με το CRD3. Δεν θέλω να επαναλάβω τα υποθέντα, αλλά προφανώ θα εξετάσουμε υποστήριξη των βασικών στοιχείων μεταρρύθμισης που έθεσαν οι G20. Έχουμε ευθύνε στην Ευρώπη να πετύχουμε στόχους όσον αφορά την ποιότητα των κεφαλαίων, να να μην υπάρξει υπερβολικό φαινόμενο μόχλευση στο σύστημα, να υπάρχει επαρκή ρευστότητα στο σύστημα και βεβαίω να μειώσουμε ναι. κυκλικά φαινόμενα. Κάτι που υπάρχει στο παρόν πλαίσιο. Για όλους τους τομείς θα πρέπει να καλυφθούν όλοι οι τομείς από την έκθεση. Είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να δω τι θα απορρέψει από τις συζητήσεις, από την ανταλλαγή απόψεων και από τις ακροάσεις και τους εμπειρογνώμονες που θα μιλήσουν διότι το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μα είναι στην πρώτη γραμμή επί του θέματος και ούτω τρόπος αντί να μένουμε πίσω και να πρέπει συνεχώς να δρούμε, αντί να δρούμε. Υποστηρίζω λοιπόν την προσέγγιση του εισηγητή. Νομίζω ότι υπάρχει μια ομοφωνία μεταξύ μας στο θέμα αυτό. Ε, θέλετε να λάβετε το λόγο και πάλι κύριε Καρά ή όχι. Η κυρία Γκέρι έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα, θα να σας ευχαριστήσω και να σταθώ σε ένα σημείο το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικό σε αυτή τη συζήτηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να κάνουμε μια σωστή αξιολόγηση αντικτύπου από τη δική μας πλευρά και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε αν αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θέλουμε να εφαρμόσουμε θα έχουν ένα ομοιόμορφο αντίκτυπο στις διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Στη συζήτηση του CRD3 είχαμε ήδη θίξει το θέμα αυτό. Εδώ θα πρέπει να δούμε όμως αν έχουμε αυστηρότερα μέτρα τα οποία θα εφαρμόσουμε. Μήπως αυτό θα οδηγήσει σε ορισμένε περιοχές της Ευρώπης, και ιδίω στην κέντρο-ανατολική Ευρώπη, θα τις οδηγήσουν σε μια μειονεκτική θέση. Είδαμε ότι η κρίση σώβησε ιδιαίτερα ισχυρά στην κέντρο-ανατολική Ευρώπη, αλλά παρόλα αυτά το τραπεζικό σύστημα μπόρεσε να επιβιώσει παρόλα αυτά. Και δεν χρειάζεται να υπάρξει επανακεφαλαιοποίηση στην Κεντροανατολική Ευρώπη όπω στη Δυτική Ευρώπη. Ήταν καλά τα αποτελέσματα των τραπεζών, αντέξανε καλά την κρίση σε σχέση με τις δυσκολίες που αντιμετωπίσανε οι τράπεζες στη Δυτική Ευρώπη που είχαν να αντιμετωπίσουν σημαντική έλλειψη ρευστότητο και δεν μπορούσαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν τα απαραίτητα δάνεια. Λοιπόν, μια αυστηροποίηση του πλαισίου θα κάνει ακόμα πιο δύσκολο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν χρηματοδότηση και αυτό θα αφορά και τις μικρομεσαίες στην Κεντροανατολική Ευρώπη. Γι' αυτό θέλω να σας ζητήσω το εξής. Αν κάνουμε μια έκθεση εκ των προτέρων αντικτύπου που θα πρέπει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να εξετάσουμε ποιες θα είναι και οι επιπτώσεις για τις διάφορες περιφερειές της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Έχουμε καθυστερήσει περίπου 40 λεπτά σε σχέση με την αρχική μας πρόβλεψη. Κύριε Κάνα, δεν θέλετε να λάβετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι το χρονοδιάγραμμα έχει αναφερθεί ήδη από τον εισηγητή και έχει διανεμηθεί σε όλους και όλοι είσαστε ενήμεροι. Μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στο σημείο υπαριθμών 5 της ημερησίας διάταξης, το θέμα των, ε, των αποδοχών των, των αμοιβών των διευθυντών των εισηγμένων στα χρηματιστήρια εταιριών και των, τις πολιτικές ε, ε, αμοιβών στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Ο κύριος Ερχαντραού είναι εισηγητής. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Οι αμοιβέ των στελεχών σε χρηματοπιστωτικές εταιρείες αυτό είναι ένα θέμα το οποίο για διαδικαστικούς λόγους δεν μπορούμε να το αναπτύξουμε σε όλη την εμβέλειά του. Επομένως θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε συγκεκριμένα θέματα. Εγώ είμαι ανοιχτό σε επικοδομητικές συζητήσεις με όλους τους σκιώδεις συζητητές και θα ήθελα φυσικά από τη δική τους πλευρά να μπορέσουμε να έχουμε σαφήνειες σε ορισμένες τροπολογίες. Εγώ ξέρω ότι μπορεί να υπάρχουν επίμαχα σημεία στα οποία θα διαφωνήσουμε, αλλά υπάρχουν απόψεις που οδηγούν σε συνένεση πέρα από τα σύνορα των πολιτικών ομάδων. Μας απασχολεί όλους το πρόβλημα πολιτικών που οδηγούν σε υπερβολική υπερβολικά επίπεδα αμοιβών. Και αυτό είναι ένα σημαντικό τμήμα μιας ευρύτερη συζήτηση η οποία είναι το πώς μια εταιρεία εισηγμένη σε χρηματιστήριο ή μια χρηματοπιστωτική εταιρεία θα πρέπει να λειτουργεί. Εγώ κατανοώ ότι η Κομισιόν θα παρουσιάσει μια πράσινη βίβλο για αυτό συγκεκριμένο το θέμα που να εστιάζει στα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου για το πώς θα λειτουργεί ο έλεγχος κινδύνων, πώς θα λειτουργεί εξωτερικός λογιστικός έλεγχος, πώς θα υπάρχει λοιπόν γενικά μια εταιρική διακυβέρνηση στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αυτό το αντιμετωπίσουμε τις επόμενες εβδομάδες και αυτό θα δώσει λαβή φυσιολογικά σε νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, κάτι το οποίο υποστηρίζω εγώ. Η χρηματοοικονομική κρίση μας έδειξε τις ε, αδυναμίες του συστήματός μας και αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε ρυθμίσεις ad hoc για να επιλύσουμε τα προβλήματα που έχουμε ενώπιόν μας. Νέες κεφαλαιοχικές απαιτήσει από τις τράπεζες, δημιουργία ενός ε, ευρωπαϊκού φορέα εποπτείας. Όλα αυτά είναι σημαντικά μέτρα σε διαφορετικό επίπεδο, αλλά πέραν αυτών θα πρέπει να πάρουμε και μέτρα που θα αφορούν την ίδια τη λειτουργία των τραπεζών. Η διαχείριση του κινδύνου σε οποιαδήποτε επιχείρηση είναι πάρα πολύ σημαντική, είτε είναι χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα, ή οποιαδήποτε εταιρεία. Μιλάμε για γενικές διαδικασίες οι οποίες θα πρέπει να ισχύουν και συμφωνίες οι οποίες θα διέπουν την πολιτική αποδοχών ώστε να μην παροτρύνουν τα στελέχη σε υπερβολικό κίνδυνο. Θέλουμε επίσης να εξασφαλίσουμε και τη διαφάνεια και όλα αυτά θα πρέπει να υπόκειται και στον έλεγχο των εποπτών και ρυθμιστών στους τομείς αυτούς. Δεν θέλω τώρα να μπω σε όλες τις λεπτομέρειες. Η Κομισιόν έχει κάνει ορισμένε ε, προτάσεις ήδη που νομίζω ότι πηγαίνουν προς σωστή, κατεύθυνση και νομίζω ότι πλησιάζουμε το σημείο που θα πρέπει να προχωρήσουμε σε κάτι συγκεκριμένο και δεσμευτικό. Εξήτασα φυσικά και την εκθέση της κυρίας Μακάρθη για τις κεφαλοχικέ απαιτήσει και περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες ιδέες η έκθεση αυτή, όπως παραδείγματος χάρη το ότι το συνολικό ε, επίπεδο αποδοχών θα πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη μορφή. Υπάρχουν στοιχεία λοιπόν τα οποία επικαλύπτονται με τη δική μου έκθεση και εγώ συμφωνώ με την κυρία Μακάρθη ότι θα πρέπει οι μέτοχοι να έχουν ένα πιο σημαντικό λόγο στο να καθορίσουν τις αποδοχές των υψηλών στελεχών σε εταιρείε που είναι εισηγμένε στο χρηματιστήριο. Θα πρέπει να υπάρξει μια επιτροπή αποδοχών στις εταιρείε αυτές και η διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου θα πρέπει να υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση των χρηματοοικονομικών εποπτών και θα πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες για να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ της διαχείρισης του κινδύνου και των λειτουργικών μονάδων σε μια επιχείρηση και αυτά πρέπει να υπόκειται λοιπόν στον έλεγχο της χρηματοοικονομικής εποπτείας. Νομίζω ότι το επίπεδο των αποδοχών θα πρέπει να καθορίζεται στο φως μακροπρόθεσμων στόχων που θα έχουν ήδη τεθεί εκ των προτέρων ώστε να μην υπάρχουν ε, δράσεις οι οποίες δεν είναι βιώσιμες. Και επίσης θα πρέπει να υπάρχει και μια λογική κατανομή των αποδοχών μέσα σε μια εταιρεία γιατί δείχνουν τα στοιχεία ότι μετά από το έτος 2000 ε, τα μπόνους, οι πρόσθετες αμοιβέ που δίνονται στα υψηλά στελέχη έχουν εκτοξευθεί στο διάστημα σε σχέση με τις αποδοχές των υπολείπων ασχολουμένων στις εταιρείε. Θα πρέπει να υπάρχουν και όρια στις ε, πληρωμές λόγω αποχώρησης και στις χρυσές χειραψίες. Δεν νομίζω ότι μπορώ να τα αναφέρω όλα αυτά. Νομίζω ότι μπορείτε απλώ να διαβάσετε το έγγραφό μου. Για να κλείσω όμως θέλω κάνω τις εξής επισημάνσεις. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία περιλαμβάνονται στην οδηγία περί κεφαλουχικής επάρκειας και αυτό είναι πολύ σημαντικό και σε ορισμένου τομεί <clears throat> τονίζω ότι ο ρόλος του χρηματοοικονομικού επόπτη θα πρέπει να είναι ισχυρότερος και αυτό πρέπει να γίνει με νομοθετική ρύθμιση. Θα ήθελα ζητήσω λοιπόν την Κομισιόν να αναλάβει τι κατάλληλε πρωτοβουλίε, ώστε να υπάρχει μια γενική εικόνα και επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο θα πρέπει να οργανώνονται οι εταιρείε σε σχέση με την πολιτική αποδοχών του. Θα πρέπει να κατονομάσουμε και να επωνυδίσουμε επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις που δεν εφαρμόζονται αυτές οι αρχές. Και τέλος, στο τέλος της εκθεσής μου, κάνω ορισμένε άλλες παρατηρήσεις, οι οποίες είναι ίσως πολιτικού χαρακτήρα περισσότερο, αλλά συνδέονται με το γενικό περιεχόμενο της έκθεσης. Παραδείγματος χάρη, ότι πρέπει να βρεθεί και κάποιος ευρωπαϊκός φόρος για τις πρόσθετες αμοιβέ, δηλαδή τα μπόνους. Αυτό θα ήταν χρήσιμο και υπάρχουν συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα τώρα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τις ε, ε, εισφορές που θα πρέπει να γίνονται σε ένα ταμείο για τις αποδοχές. Και, αποδοχές. και περιμένω και τις συμβολές των συναδέλφων. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Οι άλλοι συγγητές νομίζω θέλουν να λάβουν το λόγο. Ευχαριστώ, λέει ο Χάγκλαντ. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση. Αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να πω ότι ίσως και ένα σύμβολο στο πόσο μακριά πάει πολιτικός λαϊκισμός. Πρέπει να πετύχουμε τη σωστή ισορροπία. Πρέπει να πάρουμε μέτρα για να ρυθμίσουμε τις αμοιβέ Ίσως όμως απ' την άλλη, σαν πολιτικοί προσπαθούμε να ρυθμίσουμε πράγματα που ίσως να αφορούν τα εσωτερικά μιας εταιρείας. Δύσκολη ισορροπία λοιπόν. Και εκτιμώ την προσέγγιση του εισηγητή που συζητά το θέμα με τους κοιόδης. Είμαι σίγουρος θα καταλήξουμε σε κοινή θέση. Επί διαφόρων σημείων. Εν συντομία κάποια σχόλια, λόγω λήψης χρόνου. Εν γέννη καλή έκθεση. Εμπεριέχονται στοιχεία με τα οποία διαφωνώ. Παραδείγματο χάρη το θέμα των αποδοχών που θεωρείται ένα από τα βασικά αίτια της χρηματοπιστωτικής κρίσεως. Αυτό είναι υπερβολή, κατά την άποψή μου. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να μιλάμε για ένα ταμείο ασφάλισης, αλλά ταμείο σταθερότητας. Δεν θεωρώ ότι τα, συνδικά, τα εκπρόσωποι των συνδικάτων να πρέπει να συμμετέχουν στις συζητήσεις για την πολιτική των αποδοχών και των αμοιβών. Κατά την άποψή μου, δεν χρειάζεται να εξετάσουμε τις διαφορές μεταξύ των μεγίστων και ελαχίστων αποδοχών σε μια εταιρεία. Αυτό δεν θέμα πολιτικών, αλλά των εταιριών. Και δεν πείθομαι όσον αφορά την προσέγγιση με ποσοστά. Δηλαδή, τι ποσοστό πρέπει να καταβάλλεται σαν πόνους. Χρειάζεται ισορροπία. Αλλά η προσέγγιση με ποσοστά δεν ξέρω αν είναι σωστή. Ίσως να είναι και ο μόνος τρόπος, δεν μου πολύ αρέσει όμως. Για τις τράπεζες. Πρέπει να θυμάστε ότι όλες οι τράπεζες δεν είναι εισηγμένες εταιρείε, τουλάχιστον στις σκανδιναβικές χώρες. Πολλές τράπεζες είναι ιδρύματα και λοιπά και Οπότε δεν εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα στις σκανδιναβικές τράπεζες. Και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Δεν πιστεύω στο φόρο του μπόνους και σε αυτή την προσέγγιση. Θα υποβάλω σχετικά τροπολογίε με τα σημεία που διαφωνώ. Να δούμε που θα καταλήξουμε. Είμαι πεπισμένο ότι υπάρχουν δυνατότητες συντάξεως σωστού καλού εγγράφου που περιγράφει τις προκλήσεις πραγματικές όσον αφορά τις αμοιβέ και τις αποδοχέ, Θα πρέπει να κοιταχτούμε στον καθρέφτη και να δούμε κατά πώ θέλουμε να ρυθμίσουμε τα πράγματα για να έχουμε καλό σύστημα αμοιβή των ανθρώπων στον τομέα ή αν θέλουμε το, να το κάνουμε αυτό για λαϊκιστικούς λόγους. Κάτι που απορρέει από τη χρηματοδοτική κρίση. Χρειάζεται σωστή ισορροπία. Έχουμε δουλειά να κάνουμε. Είμαι σίγουρος ότι η τελική έκθεση θα είναι πάρα πολύ καλή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο Πασκάλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εγώ υποστηρίζω απόλυτα την γραμμή και το ύφος αυτής της έκθεσης του συναδελφού του κ. Ελχαντραουή και θα συμφωνούσα ιδιαίτερα με αυτά που είπε και ο συνάδελφός μου από τη φιλελεύθερη ομάδα ότι τα θέματα αποδοχών είναι θέματα εσωτερικά για κάθε εταιρεία. Όταν αντιμετωπίζουμε όμως ένα σύστημα για τα θέματα αυτά, το δεν είναι μονάχα το θέμα της, ε, των αποδοχών σε μία εταιρεία, σε δύο εταιρείες είναι γενικά το θέμα του πώς αποφασίζονται οι αποδοχές, πώς εξελίσσονται, με βάση ποια κριτήρια και φτάνουμε πια σε προβλήματα τα οποία είναι πολιτικού χαρακτήρα. Και όπως στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει ένα σύνολο κανόνων, είτε με συλλογικέ συμβάσεις είτε με δημόσιους νόμους που αναφέρουν τις ελάχιστες αποδοχές, τους ελάχιστους μισθούς κτλ. δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι το θέμα των αποδοχών των μισθωτών, αλλά δεν είναι πολιτικό το θέμα των αποδοχών των υψηλών στελεχών. Φυσικά δεν πρόκειται να τα θεσπίσουμε εμεί ω πολιτικοί, αλλά οι πολιτικοί πρέπει να δημιουργήσουν του κανόνε, το πολιτικό πλαίσιο που θα επιτρέψουν στου μετόχου και στα υψηλά τη στελέχη να διαπραγματευτούν τι αποδοχέ του. Επομένω, εγώ υποστηρίζω απόλυτα το πνεύμα το οποίο έχει ακολουθήσει ο εισηγητή για το θέμα αυτό και θα χαιρετήσω τις ενδεχόμενες πολιτικές προτάσεις οι οποίες μπορούν να έρθουν για το θέμα αυτό από την Κομισιόν. Τρεις παρατηρήσεις τώρα. Η πρώτη παρατήρηση αφορά το γεγονός ότι οι μέτοχοι θα πρέπει να μπορούν και να αποφασίζουν ή να απορρίπτουν το πακέτο για τις αποδοχές των υψηλών στελέχων, των διευθυντών. Αυτό νομίζω ότι είναι κανόνα ευκυβερνησία να έχουν οι μέτοχοι αυτή τη δυνατότητα και αυτό αυξάνει την διαφάνεια τέτοιου είδους αποφάσεων. Αλλά από την άλλη πλευρά, το μεταβλητό τμήμα των αποδοχών θα πρέπει να περιορίζεται και θα πρέπει να υπόκειται σε μια σειρά κριτηρίων τα οποία θα πρέπει να έχουν αντικειμενικό χαρακτήρα και χρηματοπιστωτικό χαρακτήρα πάρα πολλές φορές κάνουμε διάκριση μεταξύ ευρωπαϊκής διακυβέρνηση επιχειρήσεων και αμερικανικής διακυβέρνηση επιχειρήσεων λέγοντας ότι το ιστορικό ευρωπαϊκό μοντέλο περιλαμβάνει και άλλα κριτήρια πέραν των χρηματοπιστωτικών κριτηρίων. Έχουμε υπαναχωρήσει την τελευταία δεκαετία ίσως για τα θέματα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να επανέλθουμε και να εισαγάγουμε και άλλα κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με κοινωνική ευθύνη, με ευθύνη σε σχέση με το περιβάλλον, στην αξιολόγηση του μεταβλητού τμήματος των αμοιβών των υψηλών στελεχών. Αυτά λοιπόν είναι οι παρατηρήσει μου. Εγώ θα καταθέσω μια σειρά τροπολογιών προ την κατεύθυνση αυτή, αλλά το γενικό ύφο τη έκθεση μου φαίνεται πολύ θετικό. Ευχαριστώ, η Βίκη. Προσπαθώ να είμαι σύντομη αυτή τη φορά. Είχαμε μια συζήτηση με τον εισηγητή την προηγούμενη εβδομάδα και με πάρα πολλά από αυτά που λέει. Φυσικά όχι όλα. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονό ότι κοιτάζει το ευρύτερο θέμα τη εταιρική διακυβέρνηση και όχι μονάχα το θέμα των αμοιβών. Έχουμε μια πολύ καλή έκθεση του ΩΣΑ που εξηγεί ποια είναι η διαφορά μεταξύ του να παίρνει κανείς ρίσκα και κινδύνους που παραμένουν τα αποτελέσματά τους μέσα σε μια εταιρεία και το να παίρνει κανείς ε, κινδύνους, να αναλαμβάνει κινδύνους οι οποίοι μετά διανέμονται και πηγαίνουν κάπου όλο. Για μένα θα πρέπει να είναι η μακροχρόνια απόδοση που είναι στη βάση της, ε, των αποδοχών. Επομένως δεν πρέπει να δει κανείς μονάχα την ε, εταιρική διακυβέρνηση σε μία εταιρεία και μόνο, αλλά το ρόλο του λογιστικού ελέγχου, του εσωτερικού ελέγχου, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί σε νομικό επίπεδο. Είναι απαραίτητο λοιπόν να εξετάσουμε πολύ περισσότερο το ρόλο των, των εποπτών σε Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι μπορούν να έχουν συνεντεύξεις με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προτού αναλάβουν καθήκοντα στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών. Νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το εξετάσουμε και περισσότερο. Επίση, θα πρέπει να έχουμε την εξασφάλιση τη αναλογικότητα. Δηλαδή, υπάρχουν μερικέ φορέ μικρά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία είναι τόσο μικρά, το, ώστε δεν έχει νόημα να έχουν μια χωριστή επιτροπή για τη διαχείριση κινδύνου. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν χωριστέ ρυθμίσει για τι μικρέ εταιρείε και επίση να σκεφτούμε συνολικά και σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μονάχα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι αν εφαρμόσουμε κάποιους φόρους μονάχα στις αποδοχές στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μετακινηθούν οι εταιρείε ε, σε υπεράκτιο επίπεδο, θα γίνουν ε, υπεράκτιες εταιρείε, αλλά παραμένουν πάντα οι κίνδυνοι. Και εγώ θα παρεμβώ, θα ήθελα να παρέμβω, αλλά μάλλον δεν θα το κάνω τώρα, ίσως μπορώ να το κάνω μέσα από τροπολογίες. Θέλει να επανέλθει ο εισηγητής και να προσθέσει κάτι για να κλείσει τη συζήτηση. πάρα πολύ σύντομα. Εγώ καταγράφω όλα αυτά τα οποία λέξαν και θα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους. Εγώ είμαι έτοιμος να δω τις τροπολογίες σας και πιστεύω θα υπάρχουν πολλές ε, επικοδομητικές τροπολογίες. Μπορούμε λοιπόν όλοι μαζί να δούμε πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε. Um, uh, the... Ευχαριστώ. Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι η 10η Μαΐου και η επόμενη εξέταση τροπολογιών θα είναι την 1η Ιουνίου. Ο στόχος μας είναι να ψηφίσουμε στις 22 Ιουνίου για αυτό το θέμα. Και επομένως να έρθει αυτό το θέμα στην Ολομέλεια του Ιουλίου. Φαίνεται ότι τον Ιούλιο θα έχουμε μόνο θέματα της δικής μας Επιτροπής έτσι που πάμε. Πάμε στο σημείο 6 στην Μέση διάταξη. η ρύθμιση των ε, συναλλαγών για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εδώ έχουμε την κυρία Σουίνμπον ως εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ Χαίρομαι για την ευκαιρία να έχουμε αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή. Μα έχουν συγχαρεί πολύ από την Επιτροπή μας για την έκθεσή μου για τις πισίνες κολύμβησης και ίσως ε, αυτή είναι κάπως διαφορετική αυτή η έκθεση την οποία θα σας παρουσιάσω σήμερα ακούμε πάρα πολλά πράγματα για τις μεθόδους, τις αγορές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρξει μια γενική ρύθμιση η οποία περιλαμβάνει και την οδηγία για τα διαφημιστικά φυλάδια, για την διαφάνεια κτλ. Προβλεπόταν να υπάρχει μια εφαρμογή για όλα αυτά τον Νοέμβριο του 2007 και οι επενδυτές και οι παίκτες στην αγορά και οι ρυθμιστές Θέλω να γίνει αυτό το ταχύτερο δυνατό, αλλά τώρα φτάνουμε τα τρία χρόνια από την εφαρμογή αυτής της οδηγίας και η εισαγωγή της μεθόδου έχει συμπέσει με τη μεγαλύτερη χρηματοοικονομική αστάθεια που έχουμε γνωρίσει τα τελευταία χρόνια. Επομένως, τα δεδομένα τα οποία έχουμε συλλέξει για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής, της μέθοδ, θα έχουν επηρεαστεί από την κρίση. Ο στόχο αυτή τη νομοθεσία ήταν να αυξηθεί ο ανταγωνισμό και να εξασφαλίσουμε καλύτερη εναρμόνιση σε όλε τι ευρωπαϊκέ χρηματαγορέ. Νομίζω ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι κατανοούν ότι η κατάργηση του κανόνα της ε, συγκέντρωσης, ιδίως για τις συναλλαγές σε μετοχές, έχει οδηγήσει σε μικρότερο κόστος εκτέλεσης των ε, εντολών και έχει οδηγήσει και σε μεγαλύτερη εναρμόνιση των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών. Η έκθεση αυτή λοιπόν θα εστιάσει την προσοχή της στην υποδομή της αγοράς και ιδίως στις διάφορες πλατφόρμες εμπορίας αξιογράφων, στους κανόνες διαφάνειες πριν και μετά από μία συναλλαγή και θα αντιμετωπίσει και άλλα ε, άλλους τίτλους πέραν των τίτλων μετοχικού κεφαλαίου και ιδίως θα εξετάσει τους μηχανισμούς εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών για να υπάρχει και εκεί πλήρης προστασία των, ε, των επενδυτών. Υπάρχουν όμως και μετά την εισαγωγή της μεθόδου νέες ε, διαδικασίες συναλλαγής, ιδίως οι αλγοριθμικές ε, συναλλαγές, οι συναλλαγές υψηλής συχνότητος και έχουμε μια σειρά από συναλλαγές προϊόντων παραγόγων που απαιτούν ιδιαίτερη ρύθμιση και εξέταση. Σε αυτή τη νέα τεχνολογική εποχή λοιπόν και τη στιγμή που έχουμε μια τόσο μεγάλη ανάγκη για διαφάνεια, η εκθεσή μου θα εξαρτάσει τις λεγόμενες σκοτεινές δεξαμενές για την ε, ε, διαπραγμάτευση για την εκτέλεση μάλλον μεγάλων εντολών. Υπάρχουν ε, λοιπόν συναλλαγές και σε σκοτεινές δεξαμενές και σε φωτεινές δεξαμενές. Αυτό επηρεάζει την ε, διαφάνεια των τιμών. Και αυτή έχει επηρεάσει όλα τα, όλους τους χώρους συναλλαγών, τα λεγόμενα MTF, τις πολυμερές, πολυμερούς χώρους διαπραγμάτευσης και τα λεγόμενα SIs. Μόνο, με την, ε, μόνο στην περίπτωση των ε, εξοχρηματιστιακών συναλλαγών που γίνεται μέσω των λεγόμενων δικτύων BCN που υπήρχαν και πριν από τη μέθοδο αλλά τώρα έχουν μια απόλυτα ηλεκτρονική μορφή καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος συναλλαγών εξοχρηματιστριακά, επομένως όχι με διάφανο τρόπο. Αυτή τη στιγμή το ΣΥΖΑ συλλέχει στοιχεία για να διευκρινιστεί ο όγκος των συναλλαγών που γίνονται μέσα στο σκοτάδι σε εισαγωγικά και επομένως ποιο είναι το, το αποτέλεσμα στην αποκάλυψη των τιμών λόγω αυτού του τρόπου συναλλαγών οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν ένα πιο χωρημένο σύστημα από ό,τι στην, Ευρωπαϊκή Ένωση και ίσως μπορούμε να διδαχτούμε από τις Ηνωμένε Πολιτείε σε σχέση με τη διαφάνεια για τις σκοτεινές δεξαμενές, ιδίως σε μια εποχή που θεωρούν οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών ότι μόνο από 1% των συναλλαγών για ε, μετοχικό κεφάλαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται στο σκοτάδι, ενώ είναι 10% το αντίστοιχο ποσοστό για τις ΗΠΑ. Ίσως τα μέλη της Επιτροπής θέλουν να διαβάσουν τα έγγραφα αυτά σε σχέση με τις σκοτεινές δεξαμενές ναι. και όλους τους χώρους στους οποίους γίνονται οι λεγόμενες σκοτεινές συναλλαγές. Η έκθεση Φλούρη του 2010, την οποία ετοιμάζει η κυρία Λαγκάρτ, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Επίσης, τα έγγραφα διαβούλευσης είναι πάρα πολύ σημαντικά και η ομάδα TAB του, που δημοσίευσε μια έκθεση του Οκτωβρίου 2009 με τίτλο Σκοτεινέ συναλλαγές στην Ευρώπη» είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Λοιπόν, περιμένω τις ε, απόψεις σας σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων που πιστεύω θα βοηθήσει την εξέλιξη του εγγράφου. Thank um, Ευχαριστώ πολύ. Κάνει κάποιος άλλος, σηκώνει το χέρι του για να πάρει το λόγο. Ε? Ο κύριος Καμφέ. Όλα. Δεν σε είδα, δεν σε είδα. Όλε Σμιτ πρώτος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την εισαγωγή που έγινε. Πρώτο ερώτημα προς εσάς. Τι θέλετε να κάνουμε. Είναι καλό ή κακό για την αγορά. Ποια είναι η άποψή σας. Διότι είναι κρίσιμο αυτό να καθοριστεί. Θα μπορούσε να είναι καλό για την αγορά, για τον καθορισμό των τιμών για τη δημιουργία πιο εύρυθμης αγοράς. Προσπάθησα να μελετήσω τα έγγραφα και εγώ. Δεν ε, θεώρησα ότι θα κάνετε έκθεση για κολυμβητήρια, για πισίνες, swimming pools, αναφερθήκατε στα pools. Αν μιλάτε για σκοτάδια και διαπραγμάτευση και εμπόριο στα σκοτάδια, δημιουργείται εντύπωση ότι αυτό δεν είναι πολύ καλό. Όταν αναφερθήκαμε στο MIFID, για τις αγορές τα χρηματοδοτικά ε, μέσα, εκεί μιλούσαμε για διαφάνεια. Όλοι στην αγορά θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν τι ακριβώς ε, λαμβάνει η χώρα. Εγώ ίδιος είμαι μικροεπενδυτής και μ' αρέσει να ξέρω ότι τουλάχιστον καθημερινά δεν κάνω τι επενδύσεις μου στο σκοτάδι. Το βασικό μου επιχείρημα είναι το εξής. Αν είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αγοράς, και είναι, γιατί μεγάλωνε στην Ευρώπη και αυξανόταν, πρέπει να κάνουμε κάτι. Να πετύχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια. Χωρίς να χάσουμε ένα βασικό εργαλείο όμως για την αντιμετώπιση αυτού του είδους των συναλλαγών. Διότι είπε Σκέι ότι η νέα τεχνολογία της πληροφορικής άλλαξε την αγορά. Ήταν πιο εύκολο να αντιμετωπιστεί το θέμα όταν επολούντο ογκώδη βουνά μετοχών σε μία μέρα. Όταν γινόταν επιτόπου η συναλλαγή. Αυτό δεν γίνεται τώρα όμως. Όπως ακούς διστάζω. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε. Δεν θέλω να έχω χρηματοπιστωτικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται στο σκοτάδι. Βασικές προσπάθειες της Επιτροπής μας όπως και με τις κεφαλουχικές απαιτήσεις είναι η διαφάνεια. Τα πάντα πρέπει να γίνονται στη διαφάνεια. Και όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά θα πρέπει τουλάχιστον να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν τι γίνεται, τι συμβαίνει στην αγορά όταν ε, συμμετέχουν σε αυτές τις ευαίσθητες ε, συναλλαγές. Ευχαριστώ. Αλήν. Τι είχατε πει sensible ή sensitive εμπόριο. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την παρουσίασή της, αλλά δεν κατάλαβα τίποτε παραπάνω ως, εισηγη, ως σκιώδης, ως προς τα ερωτήματα που μας τίθενται. Και φαντάζομαι ότι αυτό συμβαίνει διότι μερικοί ανησυχούν για την έλλειψη διαφάνειας, δεν υπάρχει κανένα αξιόπιστο στοιχείο για την ύπαρξη των dark pools. πρέπει να ξέρουμε αν υπάρχουν τέτοια μέρη της αγοράς ή όχι. Σε άρθρα που διάβασα έλεγε ότι λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης, που δεν ευθύνεται αυτή βέβαια, αλλά λόγω, υπάρχει αγορά δύο ταχυτήτων και δύο πατομάτων, δύο επιπέδων. Και πάλι ευθύνεται η έλλειψη της διαφάνειας. Πρέπει να το συζητήσουμε λοιπόν και συμφωνώ με τον κύριο Σμίτ ότι πρέπει να μάθουμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι, ποιοι, ποιοι είναι, ποιος είναι ο λόγος ύπαρξης αυτών των dark pools, γιατί μερικοί λένε ότι αυξάνει, αυξάνουν τη ρευστότητα. Ότι μπορεί να υπάρχουν ωφέλη δηλαδή. Αλλά διάβασα επίσης ότι άλλοι πιστεύουν ότι πρέπει να γίνουν γνωστά όλα αυτά. Να δοθεί μεγαλύτερη δημοσιότητα. Ελπίζω να μπορέσουμε όλα αυτά να τα συζητήσουμε και να συνεννοηθούμε ως κοιόδης, Γιατί πρέπει να το τονίσουμε. Θέλω να ξέρω κατά πόσον ωφελούν την αγορά αυτές οι, αυτός ο εμπιστευτικός χαρακτήρας ορισμένων στοιχείων και να δούμε κατά πόσον δεν τη ζημιώνει μάλλον ε, λόγω της έλλειψης διαφάνειας. Γιατί γνωρίζουμε ότι είναι όλο και περισσότερες οι σκοτεινές αυτές οι συναλλαγές. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να τα μάθουμε όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να βασιστούμε στον τρόπο με τον οποίο θα απαντηθούν τα ερωτήματα αυτά. Ίσως να χρειαστεί περισσότερη έρευνα, ίσως να ζητήσουμε από την Κομισιόν να τα κοιτάξει, αλλά να μην περιοριστούμε σε μία τέρμονη τεχνική συζήτηση περί του κατά πόσον χρειάζεται προεμπορική ή μεταεμπορική διαφάνεια και τα αυτά. Να δούμε τα βασικότερα θέματα διαφάνειας. Ευχαριστώ ο Πασκάλ. Ο Πασχάλης δηλαδή. Α, ναι, συμφωνώ με την Αλίνα. Έχουμε και εδώ την ευκαιρία ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνουμε πολιτικές προτάσεις που μάλιστα να κατατεθούν πριν την τροποποίηση που ανακοίνωσε η Κομισιόν. Άρα να παίξουμε πλήρως το ρόλο μας. Καλό είναι αυτό, πολύ καλό είναι αυτό. Ορισμένοι λένε ότι υπάρχουν ωφέλη από αυτές τις σκοτεινές περιοχές, αλλά δεν ξέρουμε ε, ποια ζημία δημιουργούν. Για να μην μακρηγορήσω θα έλεγα ότι η έλλειψη διαφάνειας ε, είναι κάτι που φάνηκε ως πρόβλημα από την κρίση. Τα dark pools είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που πρέπει να γίνει γιατί όσο λιγότερη διαφάνεια υπάρχει τόσο περισσότερες δυνατότητες κερδοσκοπίας σε μικροδιαφορές στα χρηματιστήρια και άρα το trading υψηλής συχνότητας ωφελεί τελικά μόνο τους ενδιάμεσους, τους μεσάζοντες και δεν χρησιμεύει καθόλου στην πραγματική οικονομία. Απλώς ενδυναμώνει την αστάθεια και την αδιαφάνεια, η έλλειψη διαφάνειας. Και άρα οι κύριοι παράγοντες της αγοράς που ωφελούνται είναι απλώς οι traders και οι μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες. Ήδη στη Γαλλία, γιατί δεν έχω άλλα παραδείγματα, ορισμένοι διοικητές μεγάλων επιχειρήσεων εισηγμένων λένε ότι πρέπει απολύτως να αναθεωρηθεί το σύστημα αυτό γιατί ζημιώνει τις μεγάλες επιχειρήσεις που δεν ξέρουν πλέον ποιος υποβάλλει τις παραγγελίες και ποιος κάνει τι γενικότερα. Πρέπει να τους ακούσουμε και αυτούς γιατί όλος εξαιρετικός διαφέρει από την άποψη των τραπεζών που συνήθως υποστηρίζουν τις μυστικές αυτές δοσοληψίες. Όσο για το κόστος των δοσοληψιών έχει γίνει μια προσπάθεια μείωσής του αλλά πολλαπλασιάστηκαν οι χώροι στις οποίες γίνονται οι δοσοληψίες και τελικά το κόστος αναμονάδα μπορεί να μειώθηκε αλλά το γενικό κόστος εδώ και μερικά χρόνια δεν άλλαξε. Άρα δεν υπάρχει όφελος ούτε για τους επενδυτές. Μόνο για τους μεσάζοντες, πολύ περιορισμένη κατηγορία δηλαδή. Πρέπει λοιπόν να το ξαναδούμε. Δύσκολα. Η Κάθριν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και θέλω να ευχαριστήσω και το τον εισηγητή και του, την εισηγήτρια και τους κοιόδες εισηγητές. Εγώ συμφωνώ και με όλους αυτούς που λένε ότι είναι πάρα πολύ ζωτική η διαφάνεια και οι λέξεις σκοτεινές δεξαμενές είναι σαν να είναι το λόχνες με το τέρας το οποίο υποβόσκει εκεί. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με το συγκεκριμένο θέμα της, ε, του μέθοδ και της αποκάλυψης τιμής, της γνωστοποίησης μάλλον των τιμών. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, πιστεύω, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη μέσα σε αυτή την έκθεση, είτε υποστηρίζουμε αυτή την ε, διαφάνεια είτε όχι. Καταρχήν, η συγγήτρια αναφέρθηκε σε μια σειρά εγγράφων που θα ήταν πολύ χρήσιμα στην Επιτροπή μας. Μπορεί η Γραμματεία να εξασφαλίσει ότι όλοι μας θα έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα, είτε είναι με email, μέσω από μια ιστοσελίδα. Όσο πιο πολλά γνωρίσουμε, τόσο καλύτερα για το θέμα αυτό. Δεύτερον, ξέρω ότι η Κομισιόν είχε οργανώσει ένα εργαστήριο, μια, ένα σεμινάριο για τις σκοτεινές δεξαμενές. Θα ήθελα να ξέρω ποιος ήταν παρόν εκεί και ποιο ήταν το συμπέρασμα που βγήκε από αυτό το εργαστήριο. Και αυτό φυσικά συνάπτεται με την αναθεώρηση της λεγόμενης μεθόδου. Ευχαριστώ λοιπόν. Εγώ προσκαλούμε στα περισσότερα αυτά σεμινάρια, αλλά Συνήθω δεν μπορώ να το κάνω γιατί συμπίπτουν με τι συνεδριάσει τη Επιτροπή μα. Είναι πολύ δύσκολο και ενοχλητικό ότι γίνονται όλα αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα και εμεί δεν μπορούμε να είμαστε παρόντε. Αυτό το μόνο που θα ήθελα να πω, τα μόνα δύο πράγματα που θέλω να πω είναι καταρχήν σε σχέση με τον τίτλο αυτή τη έκθεση πρωτοβουλία που είναι κάπω παράξενο επειδή μιλάει για σκότεινε δεξάμενε και όλα αυτά. Εμεί το κάναμε επίτηδε, αλλά θέλαμε, δεν θέλαμε να εφεύρουμε κάτι από το μηδέν. Αλλά ο στόχος είναι να μπορέσουμε εμείς να διερευνήσουμε και ένα ευρύτερο χώρο πραγματικά τις αλγοριθμικές συναλλαγές, οι οποίες δεν είναι σκοτεινές, αλλά είναι αλγοριθμικές. Και είναι από την άλλη πλευρά, αλλά μπορούν να, να λειτουργήσουν με μεγάλη ταχύτητα και με μεγάλη συχνότητα. Είναι λοιπόν προβλήματα υποδομών, τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε στην έκθεσή μας. Γι' αυτό φέρει αυτό τον τόσο παράδοξο τίτλο και φυσικά έρχονται και άλλα πράγματα τα οποία θα παρουσιαστούν από την Κομισιόν. Θα χρειαστεί να απαντήσουμε σε όλα αυτά και να έχουμε την απαραίτητη έκθεση. Αυτή η έκθεση λοιπόν μπορεί να διευρυνθεί αν υπάρξουν και άλλα πράγματα τα οποία μας φανούν χρήσιμα. Εγώ θα ήθελα πράγματι να έχω την ευκαιρία να δω να δούμε πόσο αποτελεσματική είναι οι αποτελεσματικές οι αλγοριθμικές συναλλαγές αν βοηθούν την αγορά ή δημιουργούν προβλήματα και επίσης θα ήθελα να ξέρω πώς λειτουργούν και οι σκοτεινές δεξαμενές. Τι γίνεται όταν κανείς αρχίζει να ξεπερνάει κάποια κατόφλια. Μπορεί να μην φτάσει κανείς στο επίπεδο με το οποίο μπορεί να αγοράσει κανείς μια δεσπόζουσα θέση, αλλά μπορεί κανείς να δημιουργήσει θέσεις αγοράς εν κρυπτό με τις σκοτεινές δεξαμενές χωρίς να το καταλάβει η, η αγορά. Ακόμα και αν υπάρχει διαφάνεια εκ των υστέρων δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω τι συμβαίνει με τις ε, σκότεινες δεξαμενές. Αλλά επειδή δεν ξέρουμε ποια είναι η ημερομηνία που θα γίνει τα μεταρρύθμιση και η ανασκόπηση της μεθόδου, είμαστε λιγάκι στο σκοτάδι. Θα ήταν χρήσιμο όμως να εξετάσουμε αυτά τα θέματα, εν αναμονή και περαιτέρων πληροφοριών και η γραμματεία σίγουρα θα σας στείλει τις, τους συνδέσμους για τα διάφορα σχετικά και συναφή έγγραφα, ώστε να έχετε την ευκαιρία να τα διαβάσετε και να είστε έτοιμοι να πέσουν πολλά megabytes στο, στο email σας. Λοιπόν, ε, η συγγήτρια αν θέλει να επανέλθει και να κλείσει το θέμα αυτό. Ευχαριστώ όλους για τα σχόλιά τους. Ναι, αφορά τα σκοτεινέ τις σκοτεινές συναλλαγές, άρα είναι πολύ δύσκολα τα στοιχεία να συλλεχθούν. Είναι έγκαιρη η σύνταξη της ε, εκθέσεως, διότι οι Εθνικές Δημιστικές Αρχές το τελευταίο ενάμινο συνέλεγαν πληροφορίες για το ΣΕΖΑΡ Άρα ε, αναμένουμε πολύ σύντομα τα στοιχεία, άρα θα ξέρουμε τα στοιχεία, ποια, ποιες συναλλαγές γίνονται στην Ευρώπη στα σκοτεινά. Σε μερικές εβδομάδες θα έχουμε διαθέσιμα τα στοιχεία. Θα είναι έτοιμα τα στοιχεία όταν θα συντάσσετε έκθεση. Αν είναι κάτι καλό ή κακό, σίγουρα εσείς που ήσασταν όταν βάλαμε τις εξαιρέσεις στο MIFID θα ξέρετε ότι υπήρχαν ε, εξαιρέσεις για ομαδικές συναλλαγές, block trading, υπέροχη ορολογία, που εξυπηρετεί ένα σκοπό στην αγορά. Το θέμα είναι σε ποιο επίπεδο έχει συνέπεια όσον αφορά την διαμόρφωση τιμών και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Άρα πρέπει να εξετάσουμε εκ του σύνεγγυς τη διαφάνεια, τον, τις εξαιρέσεις από διαφάνεια των συναλλαγών πρώτου εμπορίου και τι πληροφορίες έχουμε μετά τις συναλλαγές υποβολή ε, αναφορών μπορεί να αναβληθεί για τρεις ημέρες. Δεν μου δόθηκε κανένα παράδειγμα όπου μια καθυστέρηση τριήμερη δικαιολογείται. Υπάρχουν ε, άλλοι συμμετέχοντες στην αγορά ε, που είναι πολύ, δεν θέλουν αυτή την καθυστέρηση την τριήμερη και αν έχουν δημοσιευθεί τα στοιχεία γιατί να μην δημοσιοποιούνται στο τέλος της ημέρας. Θα πρέπει να εξετάσουμε κάποια πράγματα. Τώρα, στη νέα εποχή της διαφάνειας, όπου εκεί θα πρέπει να υπάρχουν δικαιολογίες, γιατί υπάρχει αυτή η τρίμερη πρόληψη για τρίμερη καθυστέρηση. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία, καθημερινά καταφθάνουν στοιχεία, ε, έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες να επεξεργαστούμε, αλλά τις επόμενες εβδομάδες θα γίνει παρουσίαση από το Caesar στο εργαστήριο 12 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος. Άρα θα γίνει μια μεγάλη συζήτηση εκεί όπου θα έρθει το Caesar και καθένας από τους εκπροσώπους των διαφόρων χώρων που γίνονται συναλλαγές και διάφοροι φορείς θα έρθουν να παρουσιάσουν διάφορα στοιχεία, τα υπέρ και τα κατά και τα περί αλγοριθμικών συναλλαγών κλπ. Και, και οτιδήποτε άλλο πορεύσει μέχρι τότε. Η τεχνολογία πράγματι άλλαξε. Ο κόσμος προχώρησε ταχύτατα την τελευταία τριετία όσον αφορά τι ηλεκτρονικές πλατφόρμες εμπόριου και θα είναι πολύ σημαντικό να εξετάσουμε την όλη υποδομή, ούτω ώστε να αρχίσουμε να ετοιμάζουμε κάποια φιλόδοξα σχέδια σχετικά με το πώς θέλουμε να είναι αυτή η αγορά και πώς να αυξηθεί η διαφάνεια, χωρίς να είναι εις βάρος εκείνων που για οποιοδήποτε λόγο έχουν διάφορα block trading να κάνουν, θα πρέπει τα block trades να είναι εξαιρέσει ε, και να, μην υπάρει, να είναι ένα τρόπο εκφυγής. Έχουμε πολλά μαθήματα να μάθουμε θα ήθελα να έχουμε μια σφαιρική διαδικασία, να συναντώνται οι σκιώδεις αρκετά συχνά, όσο διαρκούν οι συζητήσεις και όσο καταφτάνουν στοιχεία από τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές και από το ΣΥΖΑΡ. Έχουμε αρκετά περιορισμένα χρονικά περιθώρια, αλλά θα προτείνουμε κάποιες ημερομηνίες και ας έθετε όσο το δυνατόν περισσότεροι μπορείτε σε αυτές τις συζητήσεις. Και όσο έρχονται τα στοιχεία θα ετοιμάζουμε αυτές τις συζητήσεις για να ενημερώνεστε. Ευχαριστώ για τη σκέψη που εκφράσατε. Νομίζω ότι έχουμε συντονιστεί λίγο πολύ και ευχαριστώ που μου δώσατε αυτές τις προτάσεις για να υποβάλουμε συστάσεις. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Νομίζω ότι κάναμε έναν κύκλο. Πιστέψαμε εκεί που ήμασταν. Ε, έχουμε τον Μάριο Βαλέντσα εδώ. Τη Μαρία Βαλέντσα που είναι εδώ ε, εκπρόσωπος Ευρωπαϊκή Επιτροπής θα μπορείτε να πάρετε το λόγο μετά. Εάν βέβαια δεν έχουμε χρονοτριβήσει. Μαρία λοιπόν, ε, να πεις μερικά λόγια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλωσορίζουμε αυτή την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θεωρούμε ότι ευθυγραμμίζεται με τη δική μας προσέγγιση. Αυτή η έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας και όλα αυτά που υπόθηκαν φύγουν τα θέματα που πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εξεταστούν στην αναθεώρηση του ΜΥΦΙΤ. Τώρα, όσον αφορά τα συγκεκριμένα σημεία τα οποία εφήγησαν από τους ευρωβουλευτές, θα πρέπει να πω ότι δύο ζητήματα επαναλαμβάνονται στη συζήτηση. Πρώτα απ' όλα η διαφάνεια και δεύτερον ο ανταγωνισμός και η δικαιοσύνη αν θέλετε. Αυτοί οι στόχοι είχαν καθοριστεί από το MIFID. Αυτό που θα πρέπει να γίνει 5-6 χρόνια μετά την θέτηση του ΜΥΦΙΤ είναι να δούμε κατά πόσο οι διατάξεις που έχουν θεσπιστεί μπορούν να ανταποκριθούν στους στόχους. Όλοι στην αίθουσα συμφωνούν, πιστεύω, ότι χρειαζόμαστε επαρκές επίπεδο διαφάνειας και θεμητό ανταγωνισμό. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε σε ποιο βαθμό τα dark pools βοηθούν και στη διαμόρφωση των τιμών και αποφεύγεται από σταθεροποίησης και κατά πόσο αυτά τα σκοτεινά τμήματα της αγοράς, όπως αποκληθούν, χρειάζονται περισσότερη ρύθμιση ή διαφορετικό τρόπο ρύθμισης. Άρα είμαστε συντονισμένοι. Έχουμε κοινούς στόχους και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για τα θεσμικά όργανα όσον αφορά το εργαστήριο για τη διαφάνεια. Δεν οργανώσαμε επίσημα εργαστήρια για να κάποιες άτυπες συναντήσεις όσοι ήθιστε με τους συμμετέχοντες του τομέα σε κάποιες περιπτώσεις αντί να διεξάγονται ξεχωριστές συναντήσεις με τους εκπροσώπους του τομέα, τους μαζέψαμε όλους στην ίδια αίθουσα. Όμως ε, θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία αυτή να πω ότι θα γίνουν επίσημες διαβουλεύσεις με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ελπίζουμε να είστε παρόντες. Έχουμε προγραμματίσει να οργανώσουμε δημόσια κρόαση για το MIFID ενδεχομένως το Σεπτέμβριο. Οπότε θα σας γνωστοποιήσουμε τι θα γίνει με τα χαράς να μιλήσουν και κάποιοι ευρωβουλευτές σε αυτή την δημόσια ακρόαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και δεν θες το λόγο. Καλώς ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και όπως ακούσατε το επόμενο βήμα στη διαδικασία είναι το εργαστήριο της 12ης Μαΐου. Δεν έχουμε άλλες ημερομηνίε ε, που να έχουν προταθεί. Πηγαίνουμε τώρα στο σημείο μετά της ημερήσιας διάταξης εξετάζουμε το σχέδιο εκθέσεως για, τα, για την πιστοποίηση των, των νομισμάτων του ευρώ και ποια νομίσματα ευρώ δεν πρέπει να κυκλοφορούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει ο Εδώ είμαι. Στα βουλγάρικα θα το πω γιατί είναι πολυτεχνικό το θέμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω καταρχήν να σας ευχαριστήσω για το γεγονός ότι, που, ότι με επιφορτήσατε με την έκθεση αυτή. Ο στόχος του κανονισμού αυτού είναι να θεσπίσει διαδικασίες σε σχέση με την επαλήθευση της ε, εγκυρότητος των ε, ε, κερμάτων, των κερμάτων ευρώ. Γιατί είναι μεγάλη απειλή η παραχάραξη των κερμάτων ευρώ, ιδίως για τα πιο υψηλής αξίας κέρματα. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένα πλαίσιο για την εξακρίβωση της εγκυρότητας των κερμάτων μπορεί να οδηγήσει και σε προβλήματα σε ό,τι αφορά την αναζήτηση παραχαράξεων και την πάταξή τους. Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικές μορφές και επίπεδα προστασίας των κερμάτων. Ο κανονισμός αυτός δημιουργεί ένα νομικά δεσμευτικό εργαλείο βάσει του οποίου θα μπορέσει να δημιουργηθεί ένα κοινό πλαίσιο, μια κοινή μέθοδος για τον έλεγχο των κερμάτων ευρώ που είναι σε κυκλοφορία. Το εργαλείο αυτό λοιπόν θα χρησιμοποιηθεί από τους αρμόδιους φορείς και μέσα στο πλαίσιο αυτό η πρόταση αυτή στοχεύει στο να εξασφαλίσει μια αποτελεσματική εφαρμογή σε όλη την περιοχή του ευρώ κοινών διαδικασιών για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των κερμάτων εν κυκλοφορία και των μηχανισμών ελέγχου για τις διαδικασίες αυτές. Ως εισηγητής λοιπόν εγώ συμφωνώ απόλυτα με την προσέγγιση της Κομισιόν και τις προτάσεις του Συμβουλίου. Για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το κείμενο της Κομισιόν, εμείς θα θέλαμε να θέσουμε μια σειρά από τροπολογίες στην πρόταση της Κομισιόν. Ένας από τους κύριους τρόπους, ένας από τους κύριους στόχους μάλλον του κανονισμού είναι να εξασφαλίσει ότι θα υπάρχει εγγύηση του ότι τα κέρματα τα οποία επανέρχονται στην κυκλοφορία υπόκειται σε μια διαδικασία ελέγχου και αυθεντικοποίησης. Και αυτό θα γίνεται μέσα από τα μηχανήματα τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο, στο άρθρο 5 παράγραφος 3. Μόνο τα, καλά, τα σωστά εκπαιδευμένα άτομα μπορούν να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Προφανώς αυτό θα επιφέρει και πρόσθετο κόστος για τους φορείς που κάνουν τον έλεγχο αυτό και επομένως πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να παρακρατούν ένα τέλος για την επεξεργασία, για τον έλεγχο αυτών των ε, κερμάτων. Μιλάμε για ιδρύματα γενική ένία Θα πρέπει όμως να χρησιμοποιήσουμε το εξής κείμενο. Όλες οι επιφορτισμένες αρχές θα έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν τέλη για να καλύψουν το κόστος επαλήθευσης και ελέγχου των κερμάτων. Αυτό θα πρέπει να αντικαταστήσει το κείμενο το οποίο έχει προτείνει η Κομισιόν. προτείνουμε να υπάρξει και προσθήκη μιας νέας παραγράφου, η οποία θα επιτρέψει να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος τριών ετών, ξεκινώντας την 1η Ιανουαρίου 2012. Τα κράτη-μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν ειδικέ εξαιρέσεις <clears throat> από τις ε, ρυθμίσεις της πρώτης προτάσεως για τα μηχανήματα ε, ελέγχου των κερμάτων τα οποία λειτουργούν εφόσον έχουν αποδείξει την ικανότητά τους να ανοιχνεύουν ε, κέρματα τα οποία είναι κύβδηλα ή άλλα αντικείμενα τα οποία δεν αποτελούν κέρματα. Και παραπέμπουμε στο άρθρο 5 παράγραφος 3 για τις εξελέσεις αυτές. Αυτές οι εξελέσεις θα πρέπει να εγκρίνονται μετά από διαβουλεύσεις με την CCEG. Σε σχέση με το άρθρο 6 παράγραφος 2 πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει υποχρέωση των κρατών μελών να εφαρμόσουν διαδικασίε και κατευθυντήριε γραμμέ, οι οποίε μπορούν να εξασφαλίσουν την πλήρη και επαρκή κατάρτιση των ατόμων οι οποίοι εργάζονται στη διαδικασία επαλήθευση των κερμάτων. Αυτό διευκρινίζεται και στην τροπολογία του Συμβουλίου. Αλλά εμεί έχουμε εισαγάγει μια πρόσθετη διευκρίνηση, η οποία λέει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν την εγγύηση από, τους, από τα ιδρύματα επαλήθευση των κερμάτων ότι το προσωπικό του είναι πλήρως εκπαιδευμένο για αυτό το στόχο. Επίσης τα μηχανήματα τα οποία ελέγχονται κάθε χρόνο στα κράτη-μέλη, εμείς υποστηρίζουμε το το τη συμβαστική πρόταση μηχανημάτων που καλύπτουν τα 25% των συνολικών κερμάτων που εκδίδονται από κάθε κράτος μέλος τον προηγούμενο χρόνο. Αυτό είναι ένα. ένας εφικτός αριθμός κερμάτων, όχι μόνο για τα μεγάλα κράτη-μέλη, αλλά και για τα μεγάλα κράτη-μέλη που υπάρχει μεγάλος αριθμός μηχανών επαλήθευσης. Πιστεύουμε όμως ότι αυτό το ποσοστό είναι το ελάχιστο το οποίο απαιτείται για να μπορέσει να επιτευχθεί ο κύριος στόχος της, ε, του κανονισμού, δηλαδή να προστατευτεί το ευρώ από την παραχάραξη. Εμεί έχουμε προτείνει και μια περαιτέρω διαταξή, η οποία είναι σημαντική για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ευρύτερη εμβέλεια στη διαδικασία ελέγχου των κερμάτων. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει εναλλάξ να ελέγχονται τα μηχανήματα αυτά επαλήθευσης κερμάτων. Συζητώντας με τους εμπειρογνώμονες της ΟΛΑΦ βλέπουμε ότι υπάρχει και εκπομπή αερίων τα ανοίγουν τα κουτιά με τα κερματά. Αυτό οφείλεται σε μια χημική αντίδραση η οποία ακολουθεί την χρήση διαφόρων χημικών ουσιών. Αν υπάρχει λοιπόν η λανθασμένη αναλογία χημικών ουσιών, λέει ο εισηγητής. Όταν λοιπόν υπάρχει ένας κίνδυνος για αυτούς οι οποίοι χειρίζονται τα κέρματα θα πρέπει να αυξηθεί και το τέλος, το οποίο θα είναι σε επίπεδο 20% της ονομαστικής αξίας. Αυτό το οποίο μας απασχολεί είναι να εξασφαλίσουμε και μεγαλύτερη διαφάνεια των διαδικασιών αυτών που εφαρμόζονται στην επαλήθευση των κερμάτων και προτείνουμε να υπάρξουν οι εξής προδιαγραφές. Η Κομισιόν, αφού πάρει και αναλύσει τις εκθέσεις των κρατών μελών, θα υποβάλει στην Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή μια αιτήσια έκθεση για τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με την επαλήθευση των κερμάτων ευρώ και τα κέρματα τα οποία πρέπει να τεθούν εκτός κυκλοφορίας. Εν κατακλείδη, θέλουμε να τονίσουμε ότι αυτή η έκθεση <clears throat> έχει εκπονηθεί με σεβασμό της αρχής της αναλογικότητας και της επικουρικότητας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους με τους οποίους εγώ συνεργάστηκα, εκπροσώπους του Συμβουλίου, της Κομισιόν, των πολιτικών ομάδων. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω και την ΟΛΑΦ, η οποία με βοήθησε με την εμπειρία που έχει συσσωρεύσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρέντα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι ευχαριστώ τον εισηγητή. Πάρα πολύ καλή έκθεση. Ξέρω ότι αυτό δεν είναι ένα θέμα που συζητείται εκτενώς σε πολιτικό επίπεδο, αλλά θα ήθελα να πω κάτι πάνω σε αυτό. Και έχω και κάποιες ε, προτάσεις. Έμαθα για το θέμα αυτό και έχω κάποιες ιδέες βλέπετε. Καταρχάς θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να καθορίσουμε ποιο νόμισμα δεν πρέπει να κυκλοφορεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Το κείμενο ε, θα πρέπει να είναι εύληπτο. Όταν το Συμβούλιο συζήτησε το θέμα, ο ορισμός δεν ήταν τόσο σημαντικό θέμα, αλλά για μένα είναι σημαντικό και θα πρέπει να το συζητήσουμε. Και πρέπει να μιλήσουμε και για τα μηχανήματα που ε, επιλέγουν τα νομίσματα που κυκλοφορούν. Και πότε πρέπει να αντικατασταθούν. Θα πρέπει να τεθεί προθεσμία. Διότι όποτε κάποιο σκέφτεται ένα νέο τρόπο για να παραχαράξει ένα νόμισμα, εμεί δεν μπορούμε να αγοράζουμε καινούριο μηχάνημα ή να κατασκευάζουμε νέα μηχανήματα. Διαφορετικά θα ήμασταν τελικά τακτικοί πελάτες ε, των κατασκευαστών των μηχανών και όταν θεωρείται ένα μηχάνημα ανίκανο να ξεδιαλύνει τα νομίσματα, τι το κάνεις. Δεν το πας σε ένα μαγαζί που παίρνει μηχανήματα και τα διαλύει έτσι απλώς και στο σημείο 1β λέει ότι το προσωπικό θα πρέπει να εκπαιδευμένο σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί από ένα κράτος μέλος. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να έχουμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μια τέτοια εκπαίδευση, κατάρτιση, με κοινού προσανατολισμού όσον αφορά την κατάρτιση του προσωπικού. Νομίζω ότι το κείμενο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι αρκετά καλό, αλλά σε κάποια σημεία θα προτιμούσα το κείμενο του Συμβουλίου. Και νομίζω ότι θα πρέπει πάντα να επιλέγουμε την καλύτερη διατύπωση και θα κάνω σχετικά προτάσεις εκ μέρους της πολιτικής μου ομάδας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Σίλφη. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε πάνω σε ένα θέμα που είναι και τεχνικό και στα πλαίσια των όσων συμβαίνουν και έσβησε το μικρόφωνο της ομιλήτες και δεν την ακούνε οι Ζητώ συγγνώμη, λέει Το θέμα τη εμπιστοσύνη στο κοινό νόμισμα, ακόμα και αν είναι στα κέρματα, είναι θέμα κοινού συμφέροντο. Ό,τι λοιπόν κινείται προ την ενίσχυση μια ευρωπαϊκή προσεγγίσεω, θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και από την άλλη πλευρά διερωτώ με για κάτι, ίσω να είναι ανόητο το ερώτημα, το σκέφτηκα πριν. Ποιο είναι ο ρόλο τη κεντρική, των εθνικών κεντρικών τραπεζών. Μιλάμε για τη δημιουργία θεσμών Νομίζω ότι αν δημιουργήσαμε το Ευρωπαϊκό Σύστημα των Κεντρικών Τραπεζών που συνδεόταν με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που διασυνδεόταν με τις κρατικές κεντρικές τράπεζες, είχαμε σαν στόχο τον έλεγχο των κυκλοφορούντων νομισμάτων. Ίσως να μην θεμελιώδες. Νομίζω πρώτα απ' όλα είναι ένα θέμα εμπιστοσύνης και δεύτερον να μην αυξήσουμε τον αριθμό των φορέων που παρεμβαίνουν σε αυτό το τομέα. Θα το φροντίσουμε και αυτό. Ευχαριστώ. Κρίμα λέει ο κύριος Γκίγκολτ. Και θέλω να κάνω αυτό το σχόλιο. Το βρίσκω λιγάκι ηρωνικό ότι ενώ εμείς μιλάμε για την επαλήθευση και την πιστοποίηση των κερμάτων ευρώ, στη δική μου χώρα υπάρχει μια έντονη συζήτηση για το αν ορισμένες χώρες θα πρέπει να εκδιωχθούν από τη ζώνη του ευρώ. Αυτό είναι ηρωνικό. Ακόμα και εξέχοντα μέλη αυτής της Επιτροπής που έλαβαν το λόγο στη συζήτηση που έγινε μέσα στη Γερμανία ζητούν να διαιρέσουν, θέλουν να δημιουργήσουν διαίρεση μέσα στη ζώνη του ευρώ. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα ήταν χρήσιμο να το συζητήσουμε γιατί αλλιώς η τρέχουσα συζήτηση αρχίζει να γίνεται λιγάκι ακαδημαϊκή και κενή περιεχομένου. Κάποιος άλλος θέλει να λάβει το λόγο για κέρματα, για τα κέρματα. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι μια συζήτηση για τη ζώνη του ευρώ. Φυσικά είναι έγκυρο αυτό το οποίο λέτε, ναι. Και εγώ θέλω να υποστηρίξω αυτά που είπε ο Σβέν Γκίγκολτ, λέει η κυρία Γκουλάρ. Θα δούμε λοιπόν τι ευκαιρίε έχουμε για τη συζήτηση αυτή μέσα στη μέση διαταξή μα. Ο κύριος Ξενάκης αν θέλει τώρα να λάβει το λόγο και να πει κάτι που έχουμε τώρα το χρόνο να ακούσουμε την Κομισιόν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μερικά σχόλια μονάχα. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μπίνεφ για την έκθεσή του. Η έκθεση αυτή είναι επικοδομητική και είναι αποτέλεσμα συνεργασίας. Είναι συν... επικοδομητική γιατί τα σημεία τα οποία αναφέρει ο κύριος Μπίνεφ ενισχύουν την αρχική πρόταση της Κομισιόν και είναι και μια συνεργατική πρόταση γιατί ο κύριος Μπίνεφ κατάφερε να συνενώσει πολλούς εμπειρογνώμονες στο θέμα αυτό σε μια σειρά συναντήσεων και μπόρεσε να συναθρήσει όλα τα σημαντικά στοιχεία για το θέμα αυτό και στοιχεία τα οποία έχουν απόλυτα λογικό χαρακτήρα και πρέπει να ηγερθούν από την πλευρά λοιπόν της Κομισιόν. Εγώ θα ήθελα να εκφράσω την συμφωνία μας σε γενικό επίπεδο με τις προτάσεις του κ. Μπίνεφ μπορεί τώρα να παραμείνει ένας μικρός αριθμός λεπτομεριών οι οποίες μπορούν να καλυφθούν σε τριμερές επίπεδο επίσημα ή ανεπίσημα μαζί με το Συμβούλιο και τη Γραμματεία του Συμβουλίου και την Προεδρία, την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο. Τώρα θα ήθελα να δώσω μερικές τεχνικές εξηγήσεις για τα αισθήματα τα οποία τέθηκαν από τον κύριο Μπίνεφ το τι είναι ένα, κόμμα, ένα, ένα κέρμα το οποίο δεν είναι έγκυρο. Αυτό είναι κάτι που έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε και στο παρελθόν. Θυμόμαστε ότι είχαμε μια σύσταση το Μάιο του 2007 που εξέδωσε η Κομισιόν για το θέμα αυτό, μια σύσταση της Κομισιόν, η οποία μεταξύ άλλων περιλάμβανε και κάποιο, κάποιο ορισμό για τα κέρματα τα οποία δεν ήταν έγκυρα. Τώρα, οποιοδήποτε άμεσος ορισμός για τα κέρματα αυτά δεν είναι εφικτό να δεν είναι λειτουργικός, δεν είναι εφικτό στην πράξη. Ακολουθήσαμε λοιπόν μια διαφορετική διαδικασία. Αντί να προσπαθούμε να έχουμε ένα τεχνικό ορισμό, χρησιμοποιούμε ένα λειτουργικό ορισμό. Λέγοντας, ο Άλεξ, λέγοντας ότι οποιοδήποτε κόμμα, οποιοδήποτε κέρμα το οποίο απορρίπτεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επαλήθευσης είναι άχυρο. Από την άποψη αυτή έχουμε ένα λειτουργικό ορισμό για τα άκυρα κέρματα, μόνο που δεν είναι τεχνικός, αλλά είναι λειτουργικός. Ένα δεύτερο θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε ήταν το σε ποιο σημείο, κάθε πότε μάλλον, θα πρέπει να αντικαθιστώνται οι μηχανές επαλήθευσης. Και είναι πάλι λειτουργικός ο ορισμός. Θα πρέπει να αντικαθιστούνται όταν δεν μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αυτό δεν αφορά τις ε, μηχανές μονάχα, αλλά και τα άτομα τα οποία εργάζονται με τις μηχανές αυτές. Όταν λοιπόν βρίσκουμε ή όταν βρίσκει μια εταιρεία που λειτουργεί αυτές τις μηχανές, ότι οι μηχανές της δεν μπορούν να εκτελέσουν σωστά την πιστοποίηση των κερμάτων, τότε θα πρέπει αυτές οι εταιρείε να αντικαταστήσουν τις κερματομηχανές τους. Τι κάνουμε τώρα με μια μηχανή η οποία αστοχεί. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να εξετάσουμε τώρα. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να συζητηθεί μεταξύ της αρμόδιας εταιρείας και του προμηθευτή της ε, μηχανής, του κατασκευαστή. Του... Τώρα, το τρίτο θέμα. Το τρίτο θέμα. Πολύ ενδιαφέρον. Η εκπαίδευση πρέπει να έχει πανενοσιακή διάσταση. Προς στιγμή λοιπόν λέμε και συμφωνούμε, νομίζω και τα τρία όργανα, ότι προς στιγμήν λόγω των μεγάλων διαφορών που υπάρχουν των κανόνων που ισχύουν στις χώρες μέλη πρέπει δεν πρέπει να κάνουμε υποχρεωτική την πανενοσιακή αυτή εκπαίδευση. Παρόλα αυτά, εδώ στην Κομισιόν ακόμη το σκεφτόμαστε και προετοιμάζουμε ένα ευρωπαϊκό υποχρεωτικό πρόγραμμα πιστοποίησης των εκπαιδεύσεων. Δεν λέω να είναι υποχρεωτικό, αλλά κάποια στιγμή μετά από δύο-τρία χρόνια μπορεί να επανέλθουμε, πρέπει μάλιστα να επανέλθουμε μεταξύ μεταξύ 2015 και λοιπά. Και τότε θα δούμε τη δυνατότητα να καταστεί υποχρεωτικό. Um, uh, uh, Όσο για την εμπιστοσύνη που πρέπει να έχουν οι πολίτες και οι πολίτισσες προς τα κέρματα, νομίζω ότι είναι το βασικό στοιχείο της πρότασης αυτής. Ο πολίτης πρέπει να μπορεί να έχει εμπιστοσύνη στο κέρμα που χρησιμοποιεί και η πολίτησα. Όταν έχει στα χέρια του ή στα χέρια της ένα νόμισμα και ένα χαρτονόμισμα πρέπει να γνωρίζει ότι είναι γνήσιο, ότι έχει δημιουργηθεί από έναν ενομισμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγκεκριμένο. Τώρα, ποιος είναι ο ρόλος των εθνικών κεντρικών τραπεζών. Αυτό είναι στη διακριτική ευχέρεια των κρατών. Μερικά κράτη ε, δίνουν το δικαίωμα στις κεντρικές τους τράπεζες να πιστοποιούν τη γνησιότητα των κερμάτων και των χαρτονομισμάτων άλλες. Στα νομισματοκοπία, στη Γαλλία ας πούμε, η υπεύθυνη για τη γνησιότητα των κερμάτων είναι το γαλλικό νομισματοκοπείο de Paris και εκείνοι κάνουν την εκπαίδευση κτλ. Λοιπόν, αυτά θα τα δει το κάθε κράτος. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε ένα νέο όργανο ή υπηρεσία. Νομίζω αν δεν απατώμε ότι τα είπα όλα και ότι απάντησα σε όλα τα ερωτήματα και ερωτήσεις. Δεν υπησέρχομαι βέβαια στη γενικότερη συζήτηση, δεν είναι αυτή η δουλειά μου και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες αυτές. Επανέρχομαι στον εισηγητή. Στον κυρία Θέλω να βεβαιώσω όλους τους συναδέλφους, ιδίως του Σοσιαλδημοκράτας, ότι είμαι ανοιχτό προς όλες τις συστάσεις που έγιναν και η κυρία που, που με ρώτησε για τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες θα συνεννοηθώ με τη Βουλγαρική Κεντρική Τράπεζα και θα δω τι απόψεις έχουν και θα τα μάθω όλα αυτά. Αυτά. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε. Και τώρα Έχουμε παραπάνω χρόνο 10 λεπτά. Α, παραπάνω. Ευχαριστώ τους συναδέλφους λοιπόν που υπήρξαν τόσο γρήγοροι. Τώρα πάμε στο σημείο 8. Ανάπτυξη... Α, καλά. Ε, ξέχασα να αναφέρω τη διορία κατάθεση τροπολογιών για τα κηρύματα. 10 Μαΐου, 10 Μαΐου, τον Ιούνιο, 22 Ιουνίου ψηφοφορία στην Επιτροπή και το Σεπτέμβριο στην Αλαμέλεια. Τώρα λοιπόν πάμε στο 8, το θέμα του Εδουάρδου Σικλούνα. Σχέδιο γνωμοδότηση για την ανάπτυξη του νομικού δημιουργία θέσεων εργασία στο πλαίσιο μια νέα βιώσιμη οικονομία. Ο Εδουάρδος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για γνωμοδότηση αν δεν απατώμε και βασίζεται σε, μια, ένα σχέδιο έκθεσης το σχέδιο γνωμοδότησης που μας το προώθησαν από την Επιτροπή Απασχόλησης και αφορά το δυναμικό δημιουργία θέσεων εργασία στο πλαίσιο μιας νέας βιώσιμης οικονομίας. Το σχέδιο έκθεσης βασίζεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για μία ολοκληρωμένη στρατηγική βιώσιμης οικονομίας όπου συμπεριλαμβάνονται και θέματα κλιματολογικών ενεργών, καθαρής ενέργειας, βιώσιμων μεταφορών, προστασίας του περιβάλλοντος, δημόσιας υγείας και άλλων. Και άλλα. Επίσης, η Ένωση έχει αποφασίσει να καταπολεμήσει, να συμβάλλει στον αγώνα καταπολέμησης της υπερθέρμανσης του πλανήτη, όπως ε, λέει και η περίφημη έκθεση IBCC. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι είναι οι πράσινες θέσεις εργασίας ή οι θέσεις πράσινης εργασίας και ο στενός ορισμός που δίνει η Κομισιόν είναι η ανεπτυγμένη υψηλή τεχνολογία. Απ' την άλλη βέβαια λέει επίσης ότι ακολουθεί και έναν ευρύτερο ορισμό του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας που είναι, συμπεριλαμβάνει και άλλα κριτήρια όπως την προστασία του περιβάλλοντος και οτιδήποτε αυξάνει την αποτελεσματικότητα, δηλαδή χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια, αλλά και γενικά αυξάνει την αποτελεσματικότητα. Και η έκθεση δέχεται ότι με τέτοιο ευρύ ορισμό είναι πολύ δύσκολο να μετρήσει κανείς τα πράγματα και να κάνει μία συγκεκριμένη ανάλυση. Για την ποιότητα των θέσεων εργασίας και την ισότητα των φύλων λέγονται μερικά σωστά πράγματα καθώς και τα θέματα της ευελιξίας στην αγορά εργασίας. Από την Οικονομική μας Επιτροπή νομίζω ότι πρέπει να πω ότι πρέπει να τονιστούν λίγο περισσότερο τα οικονομικές πτυχές αλλά και το, και το περιβάλλον και πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι η σφαιρική, γενική, γενικευμένη οικονομική κρίση έχει μειώσει το ρυθμό των αλλαγών στη χρησιμοποίηση πηγών ενεργείας. Αλλά αυτό δεν πρέπει, το λέω στη γνωμοδότησή μου, να εμποδίσει τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τέτοιες μειώσεις των εκπομπών διοξιδίου. Δεύτερον, μια ευρωπαϊκή στρατηγική απασχόλησης πρέπει να τονίζει τα οικονομικά στοιχεία δεδομένα που αφορούν τις κλιματολογικές αλλαγές στην ευρωπαϊκή αγορά. Και τρίτον, Ο ορισμός της πράσινης θέσης εργασίας ή της πράσινης απασχόλησης είναι κάτι που το έχει δεχτεί και το Eurostat και ο ΣΑ και έχουν δικές τους κατευθυντήριες γραμμές και αυτές πρέπει να εφαρμόσουμε και εμείς νομίζω. Ίσως και να τις ξεπεράσουμε και να συστήσουμε οι χώρες μέλη να ταξινομήσουν τις θέσεις αυτές εργασίας με διαφορετικό κώδικα νέης. Η ονοματολογία του Eurostat. Γιατί αυτή τη στιγμή οι πράσινες δουλειές είναι κατακαιρματισμένες σε διάφορους τομείς και για να τις ταυτίσουμε, να τις ταυτίσουμε λέγω, χρειάζεται χωριστή ονοματολογία και ταξινόμηση νέης για να μπορέσουμε να τις μετρήσουμε και να δούμε αν υπήρξε πρόοδος και να κάνουμε ποσοτικούς στόχους. Οι πράσινες θέσεις εργασίας δεν είναι αναγκαστικά μόνο επιστημονικές αλλά και για ανειδίκευτους εργάτες υπάρχουν τέτοιες θέσεις, πολλές δυνατότητες και πρέπει η Κομισιόν να προσέξει ιδιαίτερα τις πιο ευάλωτες ομάδες για να μην αποκλειστούν από ένα τέτοιο πρόγραμμα. Η γνωμοδότησή μου επίσης ζητάει αποτελεσματική χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη πρασίνης απασχολήσεως και βέβαια πρέπει να ετοιμαστεί και ένα πλαίσιο που να περιγράφει πώς οι κυβερνήσεις, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι θα προσαρμοστούν σε αυτές τις αλλαγές. Τέλος, να ξαναπώ για τον ορισμό. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι ορισμό θέλουμε, αλλά είναι χρήσιμος χρήσιμος ο διαχωρισμός που πρέπει να κάνουμε μεταξύ διαφόρων τομέων ανακύκλωσης, καταπολέμησης της καθαρισμού των υδάτων, χρησιμοποίηση ανανεωσίμων πηγών ενεργείας, πράσινες υπηρεσίες κλπ. Για να μην μπερδεύονται όλα μαζί στο ίδιο τσεβάλι. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ, Φίλιπ. Ναι, δουλεύει. Λοιπόν, ακόμα ζει η χώρα μου, λέω σαν Βέλγος, άρα θα ξεκολουθούμε να παραμένουμε για μερικά χρόνια. Πρώτο σχόλιο αυτό, Πρόεδρε, αν συνεχίσουμε έτσι, σύντομα ε, θα, θα αρχίσουμε να παίζουμε και χαρτιά, γιατί θα, θα έχουμε ηρεμήσει τελείως. Ευχαριστώ τον Έντ που έδωσε το σχέδιο κειμένου. Συμφωνώ με πολλά που περιέχονται. Μ' αρέσει ότι τόνισε ότι οι πράσινε απασχόληση δεν είναι μόνο για τα νεώσιμε πηγέ ενέργεια και μόνο αυτό. Επίση, εστιάστηκε στο ότι εδώ δεν μιλάμε για πτυχιούχου πανεπιστημίων. Οι περισσότερε πράσινε τη εργασία είναι για εκείνου που δεν έχουν πτυχίο πανεπιστημίου. Έχουμε έλλειψη μηχανικών κλπ. στην Ευρώπη και αυτό δεν πρέπει να το λησμονούμε. Χρειαζόμαστε και του πτυχιούχου. Τέσσερι τομεί όμω, α πάρουμε οικοδομές, κινητικότητα, ενέργεια, τρόφιμα και γεωργία. Αν τους πρασινίσουμε του τομεί, οι περισσότερε θέσεις απασχόληση θα αφορούν λιγότερο ειδικευμένε θέσεις. Και το χρειαζόμαστε. ο τόνος που θα πρέπει να δώσουμε θα είναι των δυνατοτήτων δημιουργούνται. Αυτή η πράσινη μεταμόρφωση είναι μια δυνατότητα, μια ευκαιρία για την Ευρώπη. Για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, μπορεί η οικονομία μας και η κοινωνία μας να γίνουν πιο δυνατές, όχι μόνο έναντι της αλλαγής του κλίματος, αλλά και της ω πόρων. Βελτιώνεται η αντίσταση τη οικονομία μα. κοιτάξτε τι έγινε με το ηφαίστειο την περασμένη εβδομάδα. Πώ μα αναστάτωσε. Πώς επίσης οι αλλαγές των ε, τιμών του πετρελαίου μας ε, πλήττουν. Αυτό θα πρέπει να τονιστεί. Και άλλη πτυχή. Αν μπορεί να ηγηθεί στη μεταμόρφωση αυτή η Ευρώπη είναι και μια ανταγωνιστική δυνατότητα, ευκαιρία στις παγκόσμιες αγορές. Νομίζω ότι είναι ο μόνος δρόμος ε, ούτως ώστε η βιομηχανία της Ευρώπης να ηγηθεί ξανά. Η αντίθετη όψη του νομίσματος. Αν δεν επιταχύνουμε προς αυτή την κατεύθυνση, χάνουμε την ευκαιρία και θα ακολουθούμε και δεν θα ηγούμεθα. Και αυτή δεν είναι καλή θέση. Αυτό ήταν το πρώτο. Δεύτερο. Το πώς λειτουργεί το μοντέλο της το καινοτομία στην Ευρώπη. Πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί. Το πώς θέτουμε στόχους ε, επηρεάζει το ρυθμό της μεταμόρφωσης. Θα πρέπει να θέτουμε στόχους, να μην τρεπόμαστε όσον αφορά την ε, αποδοτική χρήση των πόρων, ε, χαμηλή εκπομπή διοξιδίου του άνθρωπο κλπ. Αυτά οι στόχοι οι πρέπει να έχουν θέση. Τρίτον, αν αυτή η Επιτροπή δεν τονίζει τη σημασία τη φορολόγηση, δίνοντα μια κατεύθυνση στι επενδύσει και αμείβοντα τη σωστή συμπεριφορά και επιβάλλοντα κυρώσει στην κακή συμπεριφορά, θα χάσουν το στόχο. Αυτό πρέπει να είναι ο στόχος της Επιτροπής μας. Όλη αυτή η συζήτηση για φορολόγηση των πόρων και για ενέργεια Όλοι αυτοί είναι φόροι που με την πάροδο του χρόνου πρέπει να εξαφανιστούν. Αλλά θα πρέπει να ε, χρηματοδοτήσουν και τη μεταμόρφωση αυτή οι φόροι και να δώσουν και κίνητρα. Θα το τονίσουμε αν θέλουμε να επιταχύνουμε την μεταμόρφωση αυτή. Και τέλος, κάτι εξίσου σημαντικό, η σημασία της ποιότητας των θέσεων απασχόλησης. Αυτό έχει σχέση και με το στόχο του 2020 της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτό αφορά και τον αριθμό θέσεων απασχόληση. Θέλουμε να μειώσουμε την ανεργία από την άλλη, αν δημιουργήσουμε ως θέσεις απασχόλησης ε, και φτωχού εργαζόμενους, δεν είναι αυτός ο στόχος. Έντουαρντ είπε ο, ο συντάκτης της εκθέσεως της Επιτροπής Απασχολήσεως το τόνισε αυτό. Εγώ λέω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε την ποιότητα των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται. Περισσότερα προσόντα να απαιτούνται, λιγότερα προσόντα να απαιτούνται, αλλά ποιοτικέ θέσει απασχόληση. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία και θα προσπαθήσουμε να, προσπαθήσουμε να προσθέσουμε αξία όσο γίνεται και να μην βαρύνουμε και να φορτώνουμε την έκθεση και την κάνουμε πολυσέλιδη που κανείς δεν διαβάζει πολυσέλιδη σε εκθέσεις ούτε σε άλλους. Συγγνώμη που, που ε, έλεγα ότι ήθελες να στοιχηματίσεις. Ε, αν ήθελες να τραβήξεις κι άλλους τη συζήτηση, ο Γιώργεν Κλούτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να κάνω κάποιες κριτικές παρατηρήσεις. Εμένα με τρομάζει ότι για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως η οικονομική πλευρά της απασχόλησης δεν υπάρχει ούτε το ελάχιστο ενδιαφέρον και έχουμε μείνει τρισιοκούκος εδώ. Θέλω να ευχαριστώ τον κύριο Σκικούνα για τις ε, γενικές κατευθύνσεις της ε, Έκθεση του, της γνωμοδότησή του, μάλλον μπορώ να τι υποστηρίξω. Έχω απλώς να κάνω όμω μία ή δύο παρατηρήσει. Πρέπει να σκεφτούμε λιγάκι περισσότερο για τις ε, κοινοφελείς υπηρεσίες, ιδίω σε μια χώρα όπως η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, που έχουμε πολλές φορές ηλικιωμένα άτομα τα οποία έχουν ε, μεγάλε δυσκολίε και για τι οποίε ε, παίζουν σημαντικό ρόλο οι κοινωνικού χαρακτήρα υπηρεσίε και όπω λέγει και ο κ. Λάμπραξ, δεν πρέπει να σταθούμε μονάχα στη δημιουργία θέσεων απασχόλησεω, αλλά και στην ποιότητα των θέσεων αυτών απασχόλησεων. Φέτο είναι το έτο αγώνα κατά τη ε, ένδυα και του αποκλεισμού. Επομένω, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε να το δούμε μονάχα σε επίπεδο κοινωνικό αλλά και οικονομικό. Γι' αυτό η Google, το δικό μου κόμμα, προσπαθεί να συνδέσει τα δύο αυτά πράγματα, να δούμε λοιπόν και από οικονομική πλευρά τι γίνεται με τις θέσεις απασχόλησης και πώς μπορούμε να έχουμε θέσεις απασχόλησης οι οποίες πράγματι επιτρέπουν στα άτομα να ζουν και να ζουν με αξιοπρέπεια. Επίσης, για το πρόγραμμα του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας υπάρχει το πρόγραμμα Decent Work, αξιοπρεπής εργασία. Έχει παραπέμψει ήδη ε, ο εισηγητής στο θέμα του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας σε ό,τι αφορά τις πράσινες εργασίες, ίσως μπορεί να αναφέρει και αυτό το θέμα του Decent Work, την, το πρόγραμμα αυτό του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γιώργο. Ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και φυσικά ευχαριστώ και τον εισηγητή εδώ θα ήθελα να θίξω τα εξή. Πρώτον, ο ορισμός μιας βιώσιμης οικονομίας. Είναι δύσκολο, όπως είπαμε ήδη, να βρεθεί ένας κοινά αποδεκτός ορισμός. Στην έκθεση χρησιμοποιείται ο ορισμός του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας που είναι πολύ ευρύς. Δύσκολο να συγκριθούν τα στατιστικά στοιχεία μεταξύ τους, παραδείγματος χάριν, τι εννοούμε όταν μιλάμε για βιώσιμη οικονομία ή βιώσιμη θέση εργασίας, όσο μάλλον για πράσινη θέση εργασίας. Κατ' εμέ μπορούν να βρεθούν βιώσιμες θέσεις εργασίας σε όλους τους τομείς της οικονομίας, όποτε η θέση αυτή σχετίζεται με μια απασχόληση που να στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ας πούμε, εδώ με τα τεράστια ποσά χαρτιού που χρησιμοποιούμε δεν κάνουμε καλή χρήση της ενέργειας. Ή το ταξίδια μας στο Στρασβούργο επίσης. Εκτός όμως από το θέμα του ορισμού. Εκτός από το θέμα λέγω του ορισμού λέγω. Υπάρχει και το θέμα της φορολόγησης και της πολιτικής στήριξης αυτών των θέσεων εργασίας. Υπάρχουν αποτελέσματα ερευνών επισήμων από την Ισπανία που δείχνουν ότι μια πολιτική στήριξη μπορεί να καταλήξει σε στρέβλωση της αγοράς εργασίας και τελικά μπορεί να δώσει και λανθασμένα μηνύματα στους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες. Ίσως καλό θα ήταν να το λέει αυτό στη γνωμοδότησή μας ως πιθανό πρόβλημα. Άλλο τώρα. Άλλο τώρα λέγω. ότι οι κακές θέσεις εργασίας με ακατάλληλες συνθήκες εργασίας δηλαδή υπάρχουν και δεν έχουν όλες οι χώρες την ίδια αγορά εργασίας. Οι σκανδιναβικές ή και βόρειες λεγόμενες χώρες Είναι δύσκολο να δούμε πώς εκεί θα δημιουργηθούν βιώσιμες θέσεις εργασίας. Γιατί οι βιώσιμες θέσεις εργασίας είναι με χειρότερες συνθήκες εργασίας. talouden Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, δεν βλέπω άλλον, οπότε μπορείς να πεις κάποια πράγματα. να προσθέσω ότι θεωρώ ότι η γνωμοδότηση κατάφερε να συνοψίσει σχεδόν τα πάντα, να καλύψει σχεδόν τα πάντα. Τα κατάφερε άριστα. Μα δίνει ένα άριστο πλαίσιο για να προσθέσουμε περισσότερε λεπτομέρειε στα σημεία που ήδη επεσήμανε. Ευχαριστώ, λέει ο κ. Σικλούνα. Πράγματι. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι σχετικό αυτό που θα πω ή όχι. Εγώ ποια κατάσταση αντιμετώπισα συντάστα την ε, γνωμοδότηση. Είχα προθεσμία να υποβάλω τη γνωμοδότηση πριν δημοσιευθεί η έκθεση. Και έπρεπε να ζητήσω τουλάχιστον δύο μέρες. Να δω τουλάχιστον την έκθεση για μία μέρα πριν συντάξει τη γνωμοδότηση. Πολύ χρήσιμες οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν και σίγουρα θα καταλήξουμε σε κάποιες τροπολογίες με τις οποίες θα μπορούσα να συμφωνήσω. Σχετικά με αυτά που υπόθηκαν. Συμφωνώ ότι ο τίτλος... Α, έχασα τη σελίδα μου. Ο τίτλος είναι αρκετά φιλόδοξος. Άρα είτε θα πρέπει να έχουμε πληρέστατη έκθεση είτε όχι. Η έκθεση αναφέρεται σε κάποιες πτυχές. Εγώ θεώρησα ότι το κείμενό μας πρέπει να είναι σύντομο και περιεκτικό. συμπεριλαμβάνοντα και τι απόψει που εκφράστηκαν σήμερα. Αλλά πάντα με συνοπτικό τρόπο. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Το χρονοδιάγραμμά μα ποιο είναι. Προθεσμία υποβολή τροπολογιών 5η Μαου. Θα συζητηθούν στι 2 Ιουνίου οι τροπολογίε. Ψηφίζουμε στην Επιτροπή στι 22 Ιουνίου. Και μετά ψηφίζουμε στην καθήλια αρμόδια επιτροπή, την Επιτροπή Απασχόληση στις 14 Ιουλίου. Αυτό είναι το τελευταίο σημείο τη ημερήσια διάταξη για σήμερα. Έτσι λέει η πρόεδρο τουλάχιστον, κοιτάζοντα απελπισμένα αν έκανε λάθο ή όχι. Να σα υπενθυμίσω, σε όσου μείνατε, ότι έγιναν κάποιε μικροαλλαγέ στην ημερήσια διάταξη σε σχέση με το αρχικό κείμενο, όχι αυτό που σα σήμερα. Αύριο η βιωσιμότητα των δημοσιονομικών δεν συμπεριλαμβάνεται και η προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις γενικές κατευθείας γραμμές για την οικονομική πολιτική και, τις, και την οικονομική διακυβέρνηση θα συμπεριλαμβάνεται προς ψηφοφορία